Καλημέρα σα όλοι. μπορεί να ξεκινήσουμε το πρώτο σημείο τη μέση διάταξη. Καλώ ήρθατε στη δεύτερη ημέρα τη συνεδριάσεω μα. ορίζω οποιονδήποτε παρακολουθεί online. just to, uh, remind... Να υπενθυμίσω στα παρόντα μέλη Βλέπω ότι κραδένουν τις κάρτες ε, ψηφοφορία Θα ξεκινήσουμε στι 10 το τη μεγάλη ψηφοφορία, αφού διεξαχθεί περαιτέρω συζήτηση τη εκθεσίας Κοράτσα Μπίλ και των σχετικών τροπολογιών. Δεν έχω μάλιστα ανακοινώσει σήμερα το πρωί. To... Θα πάμε κατευθείαν λοιπόν στην έκθεση τη κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Καλωσορίζω την εισηγήτριά μα, την κυρία Ράπτη, που είναι σκιώδη εισηγήτρια, τον κύριο Λούκα που δεν είναι εδώ ακόμα, κυρία Ρούλε. Και εγώ είμαι ο άλλο σκιώδη, δύο σκιώδης παρίστανται. Και έχουμε και μια ομάδα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι εδώ. Δεν ξέρω ποιο είναι. Νίκητα Στάμπα, yes. Νικήτα Στάμπα. Την κυρία Φρανσουά Ποντσέ, την ξέρω. Και ξέρω ότι παρακολουθούσε το θέμα. Καλώ ήρθατε λοιπόν, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. χωρί να χρονοτριβήσουμε, δίνουμε το λόγο στην κυρία Κοράτσα Μπίλτ, για να μας μιλήσει για τις τροπολογίες, τις συμβαστικές τροπολογίες, για τη σημαντική έκθεσή της, έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας. Η κυρία Κοράτσα Μπίτσα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς θέλω να πω πόσο χαίρομαι για τις 132 τροπολογίες ε, που λάβαμε και τη συνεχιζόμενη εργασία για τις συμβαστικές τροπολογίες. Είχαμε δύο πολύ καλές συναντήσεις με τους Κιώδης και ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια που έλαβα κατόπιν αυτής. Ήταν μεγάλη συμμετοχή και έχω την πεποίθηση ότι μπορούμε να πετύχουμε ακόμα περισσότερες συμβαστικές τροπολογίες και προσβλέπω να ακούσω περισσότερα από τους Κιώδης και τους άλλους. Να θέσω το όλο σκηνικό, να πω περί τίνος πρόκειται. Η έκθεση αφορά τη δημιουργία ανάπτυξη και απασχόληση στην Ευρώπη. Θα ήθελα λοιπόν ζητήσω από του συναδέρφους να συνεχίσουν την επικοδομητική συνεργασία μας, να είμαστε εστιασμένοι και πειθαρχημένοι. Δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα της εσωτερικής αγοράς αυτή την έκθεση, βλέπετε. Πρόκειται περί υπηρεσιών. Θα δώσω κάποιες απαντήσεις σε δύο σημαντικότατα κατά την απόψη μου γενικά σχόλια των σκιωδών. Πρώτα απ' όλα, οι πολύ μεγάλες φιλοδοξίες και όταν μεγαλώ τα λόγια που χρησιμοποιούσαμε όσον αφορά την οδηγία περί υπηρεσιών. Κατά την άποψή μου δεν ήμασταν πολύ ε, φιλόδοξοι το 2006, αλλά τα κράτη-μέλη ήταν μινιμαλιστικά στην εφαρμογή της οδηγίας. Δεν νομίζω λοιπόν ότι εδώ ο σκοπός μας είναι να προσαρμόσουμε προς τα κάτω την προσπάθεια, αλλά αντιθέτως να αυξήσουμε τις ε, πιέσεις επί εκείνων που είναι υπεύθυνοι για την ε, εκτέλεση. Διότι η ανεξάρτητη εξολόγηση Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αφέστατη. Υπάρχει μεγάλο δυναμικό που δεν έχουμε εκμεταλλευτεί για ανάπτυξη ε, και θέσει εργασία. Δηλαδή 350 δι ευρώ για 5 με 10 χρόνια. Κάποιο μπορεί να πει τι είναι ένα εκατομμύριο πάνω, τι είναι ένα εκατομμύριο κάτω. Αλλά είναι τόσο μεγάλο ποσό όσον αφορά το ΑΕΠ που θα ερχόταν χωρίς να ξοδεύουμε και χρήματα του φορολογωμένου, που δεν μπορούμε τέτοιες εποχές κρίσης. Αξίζει λοιπόν να αναλάβουμε τις ευθύνες μας ως Κοινοβούλιο και να ασκήσουμε και άλλη πίεση στα κράτη-μέλη και γι' αυτό πιστεύω ότι η καρδιά του θέματος είναι η δυσανάλογη και υπερβολική ερμηνεία που δίνουν τα κράτη-μέλη στα άρθρα 15 και 16 όπου έχουν τη δυνατότητα εκεί να δώσουν την ερμηνεία τους. Και αν δεν ασχοληθούμε με το θέμα της κάλυψης των προβλημάτων δεν θα μπορέσουμε πραγματικά να πετύχουμε θετικά αποτελέσματα με την έκθεση τώρα που έχουμε ιστορικά ρεκόρ ανεργία στην Ευρώπη. Γι' αυτό λέω συναδέλφου το εξή. Δεν είναι ότι υπερβάλλουμε στον αφορά την οδηγία υπηρεσιών. Δεν θέλουμε να περιορίσουμε τις θεμητές, τα θεμητά δικαιώματα των κρατών μελών να νομοθετούν για τι αγορέ του. Αλλά μιλάμε για του κανονισμού, τι διατάξει που χρησιμοποιούνται για να παρεμποδίσουν του παρόχου υπηρεσιων υπηρεσιών από άλλα κράτη-μέλη χωρί να αποδεικνύουν επουδενή ότι κάτι τέτοιο ήταν αντίθετο προ το γενικό συμφέρον. Εδώ πρέπει να εστιαστούμε. Γι' αυτό με τα χαράς λέω ότι συνεργαζόμαστε στενά με το Συμβούλιο και το Συμβούλιο και εμείς συνεργαζόμαστε και ζητάμε στην έκθεση και οι δύο ζητάμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει ένα βήμα πιο πέρα από την ομάδα εργασίας του Συμβουλίου που εκεί αυτό αφορά με εσωτερική διαδικασία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει τι δεν εφαρμόζεται, αλλά μετά τα κράτη-μέλη απλώ σημειώνουν δεόντω αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο ρόλο μα είναι να ξεκινήσουμε συζήτηση, δημόσια ανοιχτή συζήτηση, ώστε οι λαοί τη Ευρώπη να γνωρίζουν πώ του στερούν θέσει απασχόληση και ποιο είναι το κόστο τη μη εφαρμογή των μέτρων και να ανέβουμε στο ύψιστο δυνατό επίπεδο. Γι' αυτό ζητάμε στην έκθεση την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματικά να καθοδηγεί στα κράτη-μέλη όσον αφορά την ερμηνεία των άρθρων 15 και 16 και ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει επίσης με περισσότερες λεπτομέρειες πού έχει γίνει η εφαρμογή λανθασμένη και ατελής. Και γι' αυτό με νοιάζει διαφορά μεταξύ εφαρμογής και πραγματικής επιβολής. επιβολής. Μιλάμε για επιβολή, υποχρεωτική εφαρμογή των μέτρων μετά από τόσα χρόνια. Όπου τόσα χρόνια δεν εφαρμοζόταν σωστά η οδηγία για τις υπηρεσίες. Γι' αυτό πρέπει να ασκούμε ισχυρέ ε, πιέσει και πολιτικό, πολιτικό στόχο πρέπει να έχουμε τη μηδενική ανοχή που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζουμε λοιπόν ότι μέχρι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όπου θα είναι στη μέση διάταξη η οδηγία περί υπηρεσιών και θέλουμε να παραμείνει στο ύψιστο δυνατό επίπεδο όσο χρειαστεί. Θέλουμε να παραμείνει και για το φθινόπωρο και ελπίζουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει συγκεκριμένες ε, προτάσεις να μας πει ακριβώς πού υπάρχουν ελλειπείς εφαρμογές και δεν πρέπει, να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ελπίζω ότι αν είμαστε συγκεκριμένοι και εστιασμένοι και επιθαρχημένοι και ενωμένοι μπορούμε να παίξουμε σημαντικό ρόλο, μπορούμε να στείλουμε το μήνυμα στα κάτι μελη να πούμε ότι είμαστε πολύ σοβαροί όσον αφορά το να είναι υπόλογα τα κάτι μελη Και ίσως θα πρέπει να κατονομάσουμε αν χρειαστεί τα κάτι μελη τα εφαρμόζουν. Και προσβλέπουμε προσπάθειε σχετικέ της Λιθουανικής Προεδρίας. Οι ήδη επαφές με την επικείμενη Προεδρία ήταν πολύ καλή. Λοιπόν, οι συνάδελφοι ανέφεραν το ότι δεν πρέπει να ξανανοίξουμε την οδηγία περιπηρεσιών. Όταν λέω ότι θα ήθελα να την τεντώσουμε λίγο, την επεκτείνουμε στο βαθμό του δυνατού, ούτω ώστε να, αντισταθ... να μπορεί να ανταποκριθεί στι μελλοντικέ προκλήσει. Δεν μιλώ για ένα άνοιγμα της ε, νομοθετικής διαδικασία. Ήταν αντιπαραγωγικό, θα εφαρμοζόταν πιο αργά τα μέτρα. Αλλά είχαμε από το 2006 και μετά ψηφική επανάσταση που δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε. Οι υπηρεσίε διαφέρουν εντελώ λόγω κινητή τηλεφωνία, διαδικτύου και των δυνατοτήτων που προσφέρουν. Μπορεί να βάζει μια μικρή κάρτα στο τηλέφωνο και να πληρώσει. Και μπορεί να κάνει δουλειά με το τηλέφωνο και την καρτούλα και να πληρώνει ε, στη μέση τη ερήμου με μια καρτούλα, με μια SIM στο τηλέφωνο, παίρνει αποδείξει και αγοράζει τη θέση. Αυτό δεν υπήρχε το 2006. Και πρέπει να είμαστε πολύ φιλόδοξοι. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί για όλου του τομεί. Έχουμε γυναίκε που έχουν τεράστιε δυνατότητε να γίνουν επιχειρηματίε. Κάτι που συμβαίνει άλλωστε να μπορούν να ανοίξουν ένα κέντρο περίθεψη των παιδιών, βρεφτικό σταθμό κλπ. σε συνολικό επίπεδο. Δεν πρέπει να περιορίζουμε το πεδίο εφαρμογή και να μην επιτρέπουμε σε όλο τον τομέα τη πρόνοια να λειτουργεί, που προσφέρει τεράστιες δυνατότητες για απασχόληση και για ανάπτυξη. Πρέπει να συμπεριληφθεί και αυτό ο τομέας. Σε αυτή τη ε, φάση θα μπορούσα να σταματήσω, προσβλέπω τα όσα θα μου πούν οι συνάδελφοι. Τώρα από πλευράς οργάνωσης θα σας μοιράσουμε ένα επίκαιρο κείμενο των συμβαστικών τροπολογιών κατά τη εβδομάδα. Σα συμπεριλάβουμε τι σημερινέ σα ε, προτάσει και εσδήποτε άλλε προτάσει θα έχετε ή σχόλια. Και θα αναφέρουμε και στην ομολογία του ΔΕΚ. Θα κάνουμε κάποιε ευκρινήσει στο κείμενο. Και προσβλέπω στη συνέχιση τη καλή συνεργασία και θα ψηφίσουμε στις 8 και 9 Ιουλίου την Εβδομάδα των Επιτροπών και στην Ολομέλεια μετά θα πάει το θέμα το Σεπτέμβριο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και προσβλέπω στο να ακούσω τα σχόλια των ε, συναδέλφων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον ενθουσιασμό με τον οποίο ηγηθήκατε αυτό του θέματος. Να ακούσουμε από τους χειώδεις συζητές μας, κυρία Ράπτη, πρώτη. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ, όπως ευχαριστώ πάρα πολύ και την Άννα Μαρία και τη Γραμματεία της Επιτροπής, γιατί με διευκολύνατε και βάλατε το θέμα αυτό για συζήτηση σήμερα πρώτο στην ημερήσια διάταξη. Και πάλι ευχαριστώ πολύ. Τις προηγούμενες εβδομάδες είχαμε συναντήσεις των σκιωδών εισηγητών και ε, πραγματικά ήταν πολύ ε, ωφέλιμες για τη δουλειά μας ε, τώρα, σχετικά με τις τροπολογίες και με τις ε, συμβιβαστικές που είχε την καλοσύνη να καταθέσει η Άννα Μαρία. Ήδη έχουμε στείλει γραπτός τις ε, παρατηρήσεις μας και άρα εδώ περιορίζομαι να πω τα ακόλουθα. Πρώτον θέλω να γίνει σαφές ότι με τις τροπολογίες τις οποίες καταθέσαμε προσπαθήσαμε να ενισχύσουμε κάποιες πτυχές της έκθεσης αυτής όπως για παράδειγμα το δικαίωμα των καταναλωτών και ο σεβασμός της εργατικής νομοθεσίας. Ζητάμε και εμείς ασφαλώς η οδηγία να εφαρμόζεται αυστηρά. Αλλά από την άλλη πλευρά είμαστε αντίθετοι στο να θεωρείται κάθε εθνική ιδιαιτερότητα ως αδικαιολόγητος φραγμός ή ως παραβίαση της οδηγίας ιδιαίτερα όταν προβλέπεται από την ίδια την οδηγία και είναι σύμφωνη με την ομολογία του δικαστηρίου της ευρωπαϊκής ένωσης. τώρα σχετικά με τις συμβιβαστικές ε, τροπολογίες ε, θέλω να πω τα εξής ε, ότι συμφωνούμε με αρκετές προτάσεις της εισηγήτριας όμως σε κάποια θέματα παρά το γεγονός ότι είμαστε κοντά ε, χρειάζεται να γίνουν ακόμη κάποιες αλλαγές κάποιες τροποποιήσεις. ένα παράδειγμα είναι ε, η παράγραφος 2 που θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να αναφέρεται πως η πρόβλεψη για ανάπτυξη μέχρι 2,6% ε, είναι μόνον από τη σωστή εφαρμογή της οδηγίας πολύ φιλόδοξη πράγμα που το αναγνωρίζει και η επιτροπή άλλα δύο βασικά σημεία, βασικά ζητήματα της οδηγίας που για, τους, για την ομάδα μας, για το S&D Group, ε, είναι βασικά, είναι θεμελιώδη. Το πρώτο θέμα είναι η αντίθεσή μας στην παρότρινση της Επιτροπής και της εισηγήτριας για την όσο το δυνατόν περισσότερο διασταλτική ερμηνεία της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Η Άννα Μαρία προηγουμένως εξέθεσε το σκεπτικό της και την ευχαριστώ γι' αυτό έτσι λοιπόν ε, εκθέτουμε και εμείς το δικό μας σκεπτικό που λέει ότι ήδη στην έκθεση επισημαίνονται τα προβλήματα ερμηνείας που έχουν παρουσιαστεί. Μια διασταλτική ερμηνεία της οδηγίας είναι πιθανόν κατά τη γνώμη μας να προκαλέσει επιπλέον θέματα ερμηνείας και νομικής ασάφειας σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κρατών μελών και των Ευρωπαίων πολιτών Επίσης, ε, νομίζω ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι διαπραγματεύσεις για να καταλήξουμε στο τωρινό κείμενο της οδηγίας ήταν πάρα πολύ έντονες. Κατόπιν όλων αυτών θεωρούμε ότι είναι αναγκαία η διαγραφή κάθε αναφοράς για διασταλτική ερμηνεία της οδηγίας. Άλλωστε γι' αυτό ακριβώς το λόγο κάνουμε και τις ενδιάμεσες αξιολογήσεις για να δούμε τι λειτουργεί, τι δεν λειτουργεί και βεβαίως να το διορθώσουμε αλλά να το διορθώσουμε ε, ε, με το σωστό τρόπο και μέσα από την προβλεπόμενη διαδικασία αναθεώρησης το δεύτερο πολύ σημαντικό ζήτημα για τους σοσιαλιστές είναι η τροπολογία 38 την οποία έχει καταθέσει η συγγήτρια με την οποία ενθαρρύνει το άνοιγμα της αγοράς των υπηρεσιών στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας. Και πάλι η Άννα Μαρία προηγουμένως ε, ανέπτυξε το σκεπτικό της. Ε, ωστόσο για μας η υπόθεση αυτή είναι κόκκινη γραμμή. Στο άρθρο 2 της οδηγίας προβλέπεται ρητά ότι εξαιρούνται οι υπηρεσίες υγείας, οι κοινωνικές υπηρεσίες σχετικά με την κοινωνική στέγαση, την παιδική μέρημνα και τη στήριξη των οικογενειών και των ατόμων που έχουν ανάγκη. Επίσης, σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 28, η οδηγία δεν θίγει κριτήρια ή όρους που θέτουν τα κράτη-μέλη για να διασφαλίσουν ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες λειτουργούν πράγματι προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και της κοινωνικής συνοχής. Άρα εμείς δεν θεωρούμε ούτε σκόπιμο ούτε χρήσιμο το να επεκτείνουμε την εφαρμογή της οδηγίας σε τομείς εκτός του πεδίου εφαρμογής και ιδιαίτερα σε ευαίσθητους τομείς όπως είναι ο τομέας της ε, κοινωνικής πρόνοιας εδώ βάζω μια τελεία και λέω βεβαίως ότι είμαστε πάντοτε στη διάθεση της εισηγήτριας για παραπέρα και συζήτηση και συνεννόηση. Ε, ευχαριστώ και πάλι και την Άννα Μαρία και τη Γραμματεία και τον Πρόεδρο για τη σημερινή διευκόλυνση. Uh, uh, Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σιλβάνα. Ο κύριος Χατζημαρκάκης, εκ μέρους ε, της, ε, του κύριου Λόκεγκάρτ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε την ε, κυρία Κοράτσα Μπίλτ, επειδή δεν ήταν εδώ, δεν εδώ ο κύριος Λόκεγκατ, ε, θα τον εκπροσωπήσω εγώ. Θα ήθελε λοιπόν να ευχαριστήσει την κυρία Κοράτσα Μπίλτ σε σχέση με τη δουλειά τη για τι συμβιβαστικέ τροπολογίε. Υπήρχαν μεγάλε πολιτικέ διαφορέ που, ανα, αντικατοπτρίζονται στι τροπολογίε και βέβαια δεν ήταν εύκολο να βρει κανεί ε, κατάλληλου συμβιβασμού. Διαβάζοντα τι τροπολογίε, είναι σαφέ ότι η, υπηρεσία, η οδηγία περί υπηρεσιών είναι ένα ένα καυτό θέμα ακόμη. Ε, έτσι όπως έχουν τα πράγματα ε, χρησιμοποιείται για να ανοίξουν πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οδηγία υπηρεσιών. Ο κύριος Λόκεργαρντ θεωρεί ότι μερικές είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής οδηγίας, αλλά ε, ως φιλελεύθερος θα έπρεπε να είναι χαρούμενος από την επιτυχία στο πλαίσιο της οδηγίας των υπηρεσιών, αλλά να μην την ξανανοίξουμε ως σύνολο. Ίσως ε, θα έπρεπε για να προχωρήσουμε να έχουμε μία προσέγγιση ανατομέα προς την ε, απελευθέρωση. Ε, η αγορά υπηρεσιών χρειάζεται βελτίωση ώστε να αποκτήσει το πλήρες δυναμικό της. έχει τις εξής ανησυχίες που τις είχε αναφέρει ήδη τον Απρίλιο. Πρώτον, πρέπει να διατηρήσουμε την πίεση στα κράτη-μέλη για να ε, συνεχίσουν τις προσπάθειές τους ε, για την εφαρμογή ε, της μηδενικής ανοχής της παραβίασης των αρχών της ελεύθερης αγοράς. Επίσης, συμφωνεί με την εισηγήτρια ότι υπάρχουν σοβαροί λόγοι δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι χρησιμοποιούν τους πρόσχημα για να μην, για να μην εφαρμόζεται η οδηγία των υπηρεσιών. Και τρίτον, πρέπει να βρούμε μία λειτουργική λύση σε σχέση με τη μη διάκριση που αναφέρεται στο άρθρο 2022. Επίσης, ε, περιμένει την υπόσχεση περί μεγαλύτερων διευκρινήσεων από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, θεωρεί όμως ότι η άποψή του αντικατοπτρίζεται συμβιβαστικές τροπολογίες και θεωρεί ότι θα, μπορέσουν, θα μπορέσουμε να ε, καταλήξουμε σύντομα σε, στο κείμενο αυτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ρούλα. Η κυρία Ρούλε, ευχαριστώ πολύ και εμείς υποστηρίζουμε την εισηγήτρια και ευχαριστούμε για την καλή συνεργασία. Αυτό που είναι και πάλι σημαντικό για μας ώστε σύντομα να συνοψίσω είναι εκείνο το ένα σημείο που θέλαμε πιο ενδυναμωμένα αυτά που έχουν επιτευχθεί να εφαρμόζονται και σε σχέση με την ε, παρότρινση και ενθάρρυνση για τα όσα έχουν επιτευχθεί μέχρι τώρα, είμαστε υπέρ του ότι οι επιπτώσεις αυτής της, υπηρεσι... της περί υπηρεσιών υπερτιμώνται. Υποστηρίζουμε λοιπόν τις τροπολογίες, συμβαστικές τροπολογίες που τα κράτη-μέλη ζητείτε να ενισχύσουν την συνιστόσα την πλευρά της εφαρμογής, της υλοποίησης. Απ' την άλλη πλευρά πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει, υπάρχει αρκετή νομική ασφάλεια και δεν είναι δυνατόν να διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής από την πίσω πόρτα. Αυτό πρέπει να αποκλείεται. Οι συμβιβασμοί οι οποίοι έχουν επιτευχθεί δεν πρέπει έμεσα να αμφισβητηθούν. Κατά τα άλλα αναμένουμε και προσβλέπουμε σε περαιτέρω καλή συνεργασία. Μία παρατήρηση όμως ακόμα, νομίζω η εισηγήτρια το προανήγγειλε προηγούμενο αυτό. Υπήρχαν κάποιες περίεργες, αξιοπερίεργες τροπολογίες που στις, ε, στους 11 και 12 λέει αντανακλώνται. Τα μέλη εδώ στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή ζητείτε μια τυποποίηση να κάνουν για τον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης μπορώ μόνο να σας πω ότι ακριβώς ε, ολοκληρώσαμε το συμβιβασμό της ε, διαπραγματεύσης για την αμοιβαία αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων. Έχουμε πολλά πετύχει λοιπόν σε αυτό το πεδίο. Δεν πρέπει σε αυτό το επίπεδο τώρα και την οδηγία περί παροχής υπηρεσιών να εντάξουμε άλλη νομοθεσία εναρμόδια για αυτήν. Αλλά το ξέρει αυτό η κυρία Κοράτσα Μπίλτ και αναμένω τις δικές της ε, τροπολογίες, τροποποιήσεις σε σχέση με τις συμβαστικές τροπολογίες. Yes, Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ με την ιδιότητά μου ως σκιώδη συγητή να πω το εξή, ε, ότι ήμουν και στο παρελθόν συγητής ε, για, τις, ε, για το θέμα για την οδηγία περί υπηρεσιών. Ευχαριστώ και εγώ την κυρία Κοράτσα Μπίλτ, γιατί έδωσε μια νέα πνοή στο όλο θέμα. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο το ότι κάποιο έρχεται με μία, βλέποντας τα πράγματα με μία ε, διαφορετική, από μια διαφορετική οπτική γωνία και τονίζει κάποιες, ε, κάποια στοιχεία, κάποιους τομείς, τους οποίους ε, ε, η εσωτερική αγορά ή υπηρεσιών μπορεί να φέρει πραγματικά αποτελέσματα. Συμφωνώ με την αλληλεπίδραση ε, του θέματος αυτού με την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Αλλά πρέπει αυτό βέβαια να το επιβάλλουμε κάπως. Το είπε η κυρία Κοράτσα Μπίλτ, νομίζω ότι και η κυρία Ρούιλε είχε τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση δεν υπάρχει απομονωμένη μόνο αυτή η ε, ε, οδηγία. Είναι τμήμα ολόκληρου πακέτου για να δουλεύει η αγορά υπηρεσιών καλύτερα και βέβαια η αμοιβαία αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, γιατί οι επαγγελματίε ε, μπορεί να φύγουν από μία χώρα και να πάνε να ασκήσουν το επάγγελμά τους κάπου αλλού, να ανοίξουν μία επιχείρηση και πρέπει να μπορούν να το κάνουν αυτό διασυνοριακά. Η ρύθμιση ε, των ε, επαγγελμάτων αυτών ε, είναι σημαντική και νομίζω ότι η οδηγία υπηρεσιών δίνει τη δυνατότητα να γίνει κάτι τέτοιο. Ένα όμως από τα κρίσιμα σημεία που παραμένουν είναι η συνεργασία μεταξύ των διοικήσεων, κάτι που τονίστηκε εδώ, γιατί ε, η εφαρμογή του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς ε, επαφίεται σε αρμόδιες αρχές που ε, πρέπει να μπορούν να ελέγχουν, τη, να ελέγχουν την δυνατότητα εγκατάσταση σε μια άλλη χώρα στις χώρες με τις οποίες συνεργάζονται. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το μελετά αυτό. Νομίζω ότι κάνει ε, μελέτες και ανατομέα, κάτι που ζήτησε και η κυρία Ράπτη, και θα ήταν χρήσιμο να ακούσουμε την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όταν θα σχολιάσει τις τροπολογίες μας. Νομίζω λοιπόν ότι όλα αυτά τα σημεία είναι σημαντικά Κάτι ακόμη το οποίο πολλές φορές το έχουμε συζητήσει εμείς εδώ στην Επιτροπή μας ε, είναι η προσέγγιση του καταναλωτή. Οι καταναλωτές από τη χώρα προέλευσης, ε, γιατί γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει καμία απέτηση να παρέχει κανείς οποιαδήποτε υπηρεσία διασυνοριακά. Είναι όμως σημαντικό αυτό και ξέρουμε ότι τα Εθνικά Κέντρα Καταναλωτών ε, ενεργούν εκ μέρου των καταναλωτών και υπάρχουν άνθρωποι που τα αναφέρουν στο Κοινοβούλιο. Οπότε είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει ε, όταν έχουμε ήδη τροπολογίες γύρω από το θέμα αυτό. Κάτι ακόμη το οποίο θα ήθελα να πω είναι η έλλειψη ε, γνώσεων των δικαιωμάτων και των επιχειρηματικών δυνατοτήτων που υπάρχουν. Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλές ε, υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών που, το γνωρίζουν, ότι είναι, που δεν γνωρίζουν ότι είναι πολύ πιο εύκολο πλέον να πάνε σε μια άλλη χώρα να εγκατασταθούν. Αυτό είναι σημαντικό για την ευρωπαϊκή οικονομία και το έχω πει πολλές φορές, ειδικότερα για παρόχους business to business. Ε, αυτή είναι η πραγματική δικαιούχη εμπροκειμένου γιατί με τη μεταφορά νέων ε, ικανοτήτων, με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε νέους τομείς, ε, με την εμπειρογνωμοσύνη που πηγαίνει από τη μία χώρα στην άλλη και δεν λέω ότι πηγαίνει προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση μόνο, αλλά το γεγονός ότι υπάρχει μια τέτοια εμπειρογνωμοσύνη που μετακινείται, ε, οποιαδήποτε συστήματα, οποιοδήποτε τομείς ε, ε, μπορούν να χρησιμεύσουν ως ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και νομίζω ότι μερικές φορές το υποτιμούμε αυτό. Θέλουμε οι συνάδελφοι στη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και τη βιομηχανική πολιτική να το λάβουν υπόψη αυτό, γιατί είναι τρόπος ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ε, ευρωπαϊκής οικονομίας και έχει δίκιο η συγχύτρια που το τονίζει αυτό. Επομένως, το πλήρες δυναμικό της αγοράς υπηρεσιών δεν είναι μόνο η αύξηση κατανάλωσης των ε, Υπηρεσιών. Είναι ένας κινητήριος μοχλός ολόκληρης οικονομίας και είναι κάτι το οποίο πρέπει να ε, το εκμεταλλευτούμε περισσότερο. Το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη έχουν επενδύσει στα ε, ενιαία σημεία επαφής ε, για να το ενθαρρύνουν αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά το πρόβλημα νομίζω που έχουμε είναι ότι οι, περισσότερες, οι περισσότεροι επιχειρηματίες δεν γνωρίζουν τις επιλογές που έχουν και δεν τις προωθούν αρκετά πρέπει να δούμε τα πιο πρόσφατα στοιχεία στα ενιαία σημεία επαφών. Υπάρχουν όλο και περισσότερα ερωτήματα που τίθενται σε σχέση με αυτό το θέμα, όμως παραμένει χαμηλός ο αριθμός. Ίσως θα έπρεπε να πιέσουμε ε, όσο το δυνατόν περισσότερο και στο υψηλότερο επίπεδο τα κράτη-μέλη, να τους πούμε ότι έχουν επενδύσει ήδη σε αυτό το θέμα είναι σαν να κάνει μια επιχείρηση, μια τεράστια επένδυση σε ένα νέο προϊόν και να ξεχνά να λέει στου καταναλωτέ ότι όντω έκανε την επένδυση αυτή και να μην είναι εκμετάλλευτο το προϊόν αυτό. Ε, στο χέρι μας λοιπόν είναι να προχωρήσουμε, να ενθαρρύνουμε ε, να προωθήσουμε τις ιδέες αυτές. Ακούσαμε λοιπόν τις απόψεις όλων των σκιωδών εισηγητών. Θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο, κύριο Σφάμπ. Θέλει κανεί άλλο ε, πριν κλείσω τον κατάλογο των ομιλητών. Έχουμε λίγο χρόνο πριν ψηφίσουμε. Κύριε Σφαμπ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δεν θα μακρηγορήσω όπω μου δίνει θεωρητικά χρόνο η μερίσια διάταξη. Το βρίσκω πολύ επικοδομητικό αυτό που είπατε εσείς από την περίοδο που είσαστε σκιώδης εισηγητής του Έλκεσης. Χαίρομαι πολύ που η συνάδελφος Κοράσα Μπίλντ αυτό το θέμα που σε πολλούς συναδέλφους είναι αϊφόρο θέμα, evergreen και για το, τα κράτη-μέλη δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλές, προσπαθεί με σθένος να το προαγάγει. Η κυρία Ρίλε ανήγγειλε, είπε πιο πριν, ότι μια δίκαια αξιολόγηση πρέπει να γίνει αυτών που, που επιτεύχθηκαν μέχρι σήμερα προτού στραφούμε σε νέα δουλειά. Ξέρω ότι μελέτες πρέπει προσεκτικά να διαβάζονται και σε σχέση με μια τέτοια εκδήλωση ένας, ε, από πλευράς καθηγητή Βόλγεμουτ ενδιαφέροντα συμπεράσματα αναφέρθηκαν. Αυτή η πρόσφατη μελέτη που λέει ότι μια ε, συνεπής εφαρμογή των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, μέσω ε, συμπλήρωσης όσον αφορά την χώρα προέλευσης που τότε δεν το είχαμε καταφέρει για την παροχή υπηρεσιών στην ΕΕ θα μπορούσε την παροχή υπηρεσιών να την αυξήσει σημαντικά 1,8% του ΑΕΠ που μέχρι σήμερα αναφέρονται σε τέτοιου είδους υπηρεσίες επιπρόσθετα 193 δισεκατομμύρια ετήσια θα μπορούσαν να παράγονται. Δηλαδή ούτε το ίμιση ούτε το μισό δεν έχουμε εκμεταλλευτεί. Ένα τρίτο περίπου, κάτι παραπάνω από το ένα τρίτο. Αν λοιπόν με σοβαρότητα στραφούμε σε αυτόν τον τομέα και δράσουμε αποτελεσματικά μπορούμε να βοηθήσουμε να συνεισφέρουμε στην ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας και αυτή τη στιγμή να προωθήσουμε πολλά πράγματα τα οποία εξετάζουν για τη διάσωση του ευρώ οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Νομίζω ότι επιτυχώς με 11 άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, μια τέτοια πρωτοβουλία έχει ξεκινήσει. Νομίζω και η Σουηδία συμμετέχει στην ευρωπαϊκή ε, εσωτερική αγορά να προχωρήσουμε. Και αυτή τη μελέτη που έχουμε που υπολόγισε τι θα είχε ως αποτέλεσμα αυτών, της υπογραφής αυτών και ένταξης αυτών των κρατών Ηνωμένου Βασιλείου και Σουηδίας. Αν άνοιγαν λοιπόν οι αγορές αυτών των 12 κρατών μελών και χρησιμοποιούσαμε το δυναμικό μας θα καταλήγαμε στα 147 δισεκατομμύρια ετήσια όσον αφορά την πρόσθετη αξία. Είναι δίκαιο λοιπόν ε, να είμαστε, ας το πω ε, για εκείνους που ήταν υπερβολικά επιφυλακτικοί να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα και να δούμε τα σημαντικά ωφέλη που συνεπάγεται αυτή η πρωτοβουλία. Τέλος, τέλος, πιστεύω ότι έχει δίκιο η κυρία Ρούιλε τα όσα έχουμε επιτύχει πρέπει να είναι σεβαστά και να τηρούνται. Παραμένει βέβαια μεγάλη πορεία που πρέπει να καλύψουμε ακόμα, αν θέλουμε όλο το δυναμικό να το εκμεταλλευτούμε, αυτό που μας προσφέρει η εσωτερική αγορά δηλαδή. Και φυσικά υπάρχουν θεμητές, ε, θεμητοί φόβοι σε κάποια κράτη-μέλη και για κάποιες δραστηριότητες στα κράτη-μέλη. Στο τέλος τέλος όμως η οικονομική μας κατάσταση θα οδηγούσε μακροπρόθεσμα να επωφεληθούμε όλοι και γι' αυτό είναι χρήσιμο αυτό που είπε η κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Μόνο αν με σθένος δώσουμε συνέχεια στο θέμα μπορούμε να πετύχουμε κάποιες αλλαγές. Η έκθεση πρωτοβουλίας της νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει να κάνουμε ένα βήμα προς τα εμπρός. Ευχαριστώ. Um, Υπάρχει άλλος που να θέλει να πάρει το λόγο. Εν τη αυτή η περιπτώση θα ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν έχει να μας πει κάτι ίσως να με ενημερώσει και για κάποιες δικές τους πρωτοβουλίες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λίγη ησυχία για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακαλώ λέει ο Πρόεδρος. Είχαμε τη δυνατότητα να το επαναλάβουμε αλλά το ξαναλέμε. Είναι πρόσδεκτη αυτή η πρωτοβουλία και η συζήτηση επακολουθεί διότι πράγματι πιστεύουμε ότι η πλήρης εφαρμογή της οδηγίας υπηρεσιών είναι κάτι σημαντικό. Ε, εμπεριέχει πολλές δυνατότητες και η πλήρης εφαρμογή της οδηγίας απαιτεί σημαντική πολιτική υποστήριξη και είναι πολύ σημαντικό βήμα αυτή η έκθεση πιστεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Επί του παρόντος επεξεργαζόμεθα ε, την ε, εξέταση του κειμένου από διάφορους ομοτήμους οπότε αυτό θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε το πώς τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν την οδηγία και πιο συγκεκριμένα την αρχή της αναλογικότητας η ε, οποία αναφέρεται στην έκθεση και σωστά διότι πράγματι πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει περαιτέρω δουλειά στον τομέα αυτό και αυτό συζητούμε με τα κράτη-μέλη. Καλωσορίζουμε και αυτό που αναφέρεται για την ε, ανάγκη για περαιτέρω βεστιτοποίηση και τα σημεία επαφής, όλες οι πληροφορίες που είχαμε από επαφές μας και στα πλαίσια της υψηλής ομάδας περιπηρεσιών που δημιουργήθηκε πρόσφατα, οι πληροφορίες αυτό μας λένε επιχειρήσεις έλεγαν ότι χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την κατάσταση, το νομικό πλαίσιο. Τους χρειάζεται κάτι τέτοιο για να μπορέσουν να κινηθούν ε, από πλευρά δραστηριοτήτων σε διασυνοριακό επίπεδο. Πράγματι, έχουν γίνει πολλές επενδύσεις όσον αφορά τα ενιαία σημεία επαφής και απ' την άλλη υπάρχει μεγάλη ανάγκη ε, για πληροφορίες από πλευράς επιχειρήσεων. Άρα θα πρέπει η προσφορά και η ζήτηση να έρθουν σε επαφή. Χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία αυτό το θέμα των ενιών σημείων επαφής. Υπάρχει μια χάρτα που ενεκρίθη πρόσφατα στο Συμβούλιο και είναι κάτι που μας δίνει στέρεο έδαφος για να προχωρήσουμε. Για να προχωρήσουμε στα σημεία ενιαίας επαφής δεύτερης γενιά. Πιθανότατα θα υπάρξει κάποια άλλη πρωτοβουλία επί Λιθουανικής Προεδρίας όσον αφορά αυτά τα σημεία επαφής. Τέλος, άρθρο 20. Προετοιμάζουμε προσανατολισμούς, κατευθυντήριες γραμμές που ανακοινώθηκαν. Θέλουμε να ετοιμάσουμε πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές βάσει θετικών εμπειριών, επιχειρήσεων, καταναλωτών, ε, από πλευρά ενώσεω καταναλωτών, διότι ισχυρότατο μηχανισμό εφαρμογή του άρθρου 20 είναι η διαφάνεια. Ο κόσμο πρέπει να γνωρίζει τι διαφορέ που υπάρχουν όσον αφορά τι τιμέ. Και θα μπορέσουν να προσαρμοστούν έτσι οι επιχειρήσει και να έχουν μια συμπεριφορά που είναι πιο φιλική για την εσωτερική αγορά και κάτι που λησμόνησα. Είναι σημαντική η διάδραση μεταξύ διαφόρων τομέων της οδηγίας υπηρεσιών και άλλων νομοθετημάτων αναφέρθηκε ο σημαντικό στοιχείο θα υποβληθεί η σχετική ανακοίνωση για τα επαγγελματικά προσόντα και για την οδηγία τη σχετική για την αμοιβαία αξιολόγηση του σχετικό σύστημα και μαζί με την ανακοίνωση θα υποβληθεί και έγγραφο ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την νομική μορφή για τις ε, κατοχή μετοχών κλπ. Άρα μαζί θα δώσουμε και τον ημερωτικό έγγραφο που θα συνοδεύει αυτή την ε, ανακοίνωση. Ευχαριστώ πολύ. Η έκθεση ήρθε σε σωστή στιγμή σε σχέση με αυτά που κάνετε εσείς, λέει ο Πρόεδρος, και θα τροφοδοτήσει και τη συζήτηση στην Ολομέλεια, αν καταφέρουμε να αναβαθμίσουμε τη συζήτηση από αυτού του σημείου. Ίσως θα το λάβουμε αυτό υπόψη, διότι υπάρχει γενικότερο συμφέρον. Η ε, κυρία Κοράτσα Μπίλτ, να σας δώσω το λόγο για να συνοψίσετε όσα ακούσατε. Είμαστε καθοδόν προς ψηφοφορία στις 8 και 9 Ιουλίου, έτσι. Επιβεβαίωση είναι αυτή. 9 Ιουλίου. Ευχαριστώ λέει κύριο Κοράτσα Μπίλτ. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους και τους κοιόδης όλος ιδιαίτερος. Ήταν πολύ επικοδομητικά τα σχόλιά τους και έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε μαζί. Καταρχάς, πρέπει να αναγνωρίσουμε τη θαυμάσια δουλειά της κυρίας Γκέπαρτ, του Μάλκομ Χάρμπορ και άλλων δουλειά που έκαναν επί σειρά ετών για να παραμείνει η προσοχή σε αυτό το θέμα και να εφαρμοστούν τα μέτρα. Πολλά συνέβησαν και συμβαίνουν. Ποια είναι η προστιθέμενη αξία. Η προστιθέμενη αξία είναι να προχωρήσουμε προς τα μπρος και να οικοδομήσουμε στα επιτευθέντα αντί να επαναλαμβάνουμε τα ίδια. Σίγουρα πολλά έχουν επιτευχθεί και αυτό πρέπει να αναγνωριστεί. Και ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους οι οποίοι ενεπλάξαν στην προσπάθεια. Ευχαριστώ για την τροπολογία για τους καταναλωτές ήταν πολύ καλή και ακρόαση όπου οι εκπρόσωποι των, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτών έθεσε διάφορα θέματα όσον αφορά τη διάκριση λόγω επικότητας και διαμονής που υπήρξαν διακρίσεις και έχουν βρεθεί θετικές λύσεις. Θα υποστηρίξω λοιπόν τις τροπολογίες που αφορούν τους καταναλωτές και αυτή τη διάσταση της οδηγίας υπηρεσιών, πάρα πολύ σημαντικό. Όπως είπε και ο Μάλκολμ, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε πλήρως την υποχρέωση προς πώληση. Είναι ελεύθερες αυτές οι συμβασιακές σχέσεις. Αυτή, τη την αγορά θέλουμε. Να διευκρινίσω και κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν ο στόχος είναι φιλόδοξος ή όχι. 2,6% αύξηση του ΑΕΠ. Το πολιτικό μήνυμα είναι ότι υπάρχει τεράστιο δυναμικό χρησιμοποιητό που δεν κοστίζει τίποτα στον φορολογούμενο για να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης και ε, ανάπτυξη. Δεν θα συζητήσω τώρα το ποσοστό, μια ποσοστία μονάδα πάνω, μια κάτω. Πιο συγκεκριμένα, ερμηνεία της οδηγίας υπηρεσιών. Δεν προτίθεμαι να ξαναανοίξω το θέμα ή να προσθέσω νέους τομείς ή να ξανανοίξω κατά τρόπο μια νομοθετική διαδικασία πρέπει να δώσουμε πλήρη ερμηνεία στην οδηγία, να υποστηρίξουμε τη διασυνεργειακή εγκατάσταση που ήδη έχει δρομολογηθεί. Μπορώ να τα αναδιατυπώσω που να αναφέρει να, ότι γίνεται απόλυτα σεβαστό το άρθρο Ήδη χορηγούνται υπηρεσίε στον τομέα τη φροντίδα και τη πρόνοια συνοριακά. Δεν πρέπει να το σταματήσουμε αυτό. Αν δημιουργούν νέε απασχόληση, αν δημιουργούνται νέε εταιρείε, αν δίνονται δυνατότητε σε περισσότερε γυναίκε να δουλέψουν. θα πρέπει να, αν δεν προωθήσουμε την ε, καινοτομία, δεν πρέπει να την μπλοκάρουμε. Και η ψηφιακή τεχνολογία προοδεύει με αστραπιούς ρυθμούς. Θα αλλάξει εντελώ τον τρόπο πωλήσεων υπηρεσιών και προϊόντων. Και όπως είπε και πολύ καλά ο Μάλκομ, όλα αυτά πάνε μαζί. Δεν είναι η βιομηχανία κατά υπηρεσιών και το αντίστροφο. Το μέλλον της οικονομίας είναι ολοκληρωμένη οικονομία και ο τομέας των υπηρεσιών και των αγαθών είναι ένα κομμάτι της λύση να έχουμε ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, θα λειτουργεί εύρυθμα. Και ευχαριστώ κύριε Ρούλε που υπενθυμίσατε το... και τη σχέση με την οδηγία για τα επαγγελματικά προσόντα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ζητήσαμε στους συναδέλφους να ευκρινίσουν την ορολογία. Είναι σημαντικότατο αυτό. Πρέπει να διευκολύνουμε στο μέτρο του δυνατού την αλληλεπίδραση μεταξύ σημαντικών νομοθεσιών και να αποφύγουμε τις φαιές ζώνες. Αυτό θα ληφθεί υπόψη σίγουρα. Το συζητήσαμε και προηγουμένως. Ευχαριστώ τους συναδέλφους της ΑΛΔΕ για την υποστήριξή τους και μας υπενθύμισαν ότι βασικό θέμα είναι το κοινό συμφέρον που είναι βασικό στοιχείο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είπε ότι ετοιμάζει κατευθυντήριες γραμμές πρακτικής φύσεως για τα κράτη-μέλη πάνω σε αυτόν τον τομέα και την ευχαριστούμε γι' αυτό. Και το άλλο αυτό που έθιξε ο Ανδρέας Σφάμπ μια, την έκθεση α, περί ανοιχτής Ευρώπης και αυτό είναι συναγερμός για μας διότι στα κράτη-μέλη συζητείται διευρυμένη, αυξημένη συνεργασία και υπάρχουν σοβαρές δυνατότητες εκεί και είναι μία από τις συστάσεις εκθέσεως. Δηλαδή κάποια κράτη-μέλη θα αισθανθούν ότι θέλουν να προχωρήσουν διότι τα ωφέλη που χάνουν όσον αφορά ανάπτυξη και απασχόληση είναι πάρα πολύ μεγάλα για να περιμένουν τους άλλους. Κατά την άποψή μου το Κοινοβούλιο υπέχει καθήκον να κρατήσει την Ευρώπη ενωμένη, 27 συν 1, να δείξει τα ωφέλη μιας ολοκληρωμένης ενωμένης ανοιχτής εσωτερικής αγοράς και αν έχουμε 12 κράτη-μέλη που προχωρούν με τη διευρυμένη, με την αυξημένη συνεργασία, αυτό θα αυξήσει τον κατακαιρματισμό και θα αυξηθεί ο κίνδυνος να έχουμε Ευρώπη δύο ταχυτήτων και το οικονομικό χάσμα που είναι ένα από τα βασικά μας προβλήματα στην Ευρώπη θα αυξηθεί. Γι' αυτό θα ήθελα να έρθω σε αυτά που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τη σαφή γραμμή που παρουσιάστηκε για μεγιστοποίηση των οικονομικών ε, ωφελών, ε, να δούμε άξιο του οικονομικού ωφέλους μάλλον, συγγνώμη, να μην στερούμε θέσει επασχόληση από του Ευρωπαίου πολίτε. Και αυτό που είπε, Μάλκομ, για ευαισθητοποίηση, για ενημέρωση, είναι σημαντικότατο και καλωσορίζω αυτή την χάρτα που αναφέρθηκε για τα ε, μοναδικά σημεία επαφής δεύτερης γενιάς που ανέφερε μάλλον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οθέτησε το Συμβούλιο πρέπει να συνεργαστούμε για να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση για το Solvit, αυτά τα σημεία επαφής και πληροφορίες και για το σύστημα πληροφοριών εσωτερικής αγοράς. Ίσως θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην εβδομάδα της ενιαίας αγοράς και άλλες δραστηριότητες που ετοιμάζουμε μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αύξηση τη ευαισθητοποίηση για τι δυνατότητε που έχουν επιχειρήσει να λειτουργούν και να εγκαθίστανται σε άλλα κράτη-μέλη και για του καταναλωτέ να απολαμβάνουν την ενιαία αγορά. Κύριε Πρόεδρε, μετακινούμενοι προς το τελικό στάδιο των συμβαστικών τροπολογιών εν ώψη της ψηφοφορίας, ζητώ από τους συναδέλφους να συνεργαστούμε, να μην αποδυναμώσουμε το βασικό μήνυμα που είναι η πλήρης εφαρμογή από όλα τα κράτη-μέλη και στο ύψιστο ε, ε, πολιτικό επίπεδο να υπάρξει προσπάθεια ούτως ώστε πράγματι να εφαρμοστεί αυτή η προσπάθεια για την εκμετάλλευση ε, όλων των δυνατοτήτων απασχόλησης που προσφέρει η νέα αγορά. Αυτά και ευχαριστώ τους συναδέλφους για την προσοχή τους. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, που ηγηθήκατε σε αυτό το θέμα. Θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή 9 Ιουλίου. Παρακαλώ, λίγη ησυχία αν έχει την καλοσύνη και θέλουμε να πάμε στην Ολομέλη του Σεπτεμβρίου και θα ζητήσουμε τις πολιτικές ομάδες να δούμε μήπως μπορούμε να έχουμε και άλλη συζήτηση ενδελεχέστερη για το θέμα αυτό. Κυρία Κοράτσα Μπίλτ, αν εσείς και η ομάδα σας μαζί με τις άλλες ομάδες κινηθείτε ίσως να ζητήσουμε κάτι πιο σημαντικό, πιο σημαντική συζήτηση από ότι μια απλή συζήτηση στα πλαίσια εκθέσεως ιδίας πρωτοβουλίας. Ίσως μπορείτε να το προσπαθήσετε. Να ζητήσω και από την κυρία Ράπτη που έφυγε νομίζω και από άλλους να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Καλώ, θα ψηφίσουμε τώρα. Αν μπορείτε να καθίσετε και να ησυχάσετε, θα χρησιμοποιήσουμε τις κάρτες ψηφοφορίας. Να είστε σίγουροι ότι είναι στη θέση τους και ότι λειτουργούν οι κάρτες. Θα υπάρξουν, θα υπάρξουν κάποιες επίμαχες ψηφοφορίες, έχουμε πολλές να κάνουμε. Αν είστε στη θέση σας μπορούμε να ξεκινήσουμε.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 I'll take my first of all. Λοιπόν, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι που ήρθατε για τις ψηφοφορίες όλοι. Θα ήθελα να προτείνω μια μικρή αλλαγή στη σειρά των ψηφοφοριών. Δεν ακούσατε ακόμα αυτό το οποίο θέλω να σας πω. Μην αρνείστε πρωτού ακούσετε κύριε Σμιτ και εσείς. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι όλο και όλο να προχωρήσουμε σε σχέση με το πρώτο θέμα την εξέταση της δικής μου έκθεσης ώστε να υπάρξει έγκριση από πλευρά σας για την έκβαση του τριμερού διαλόγου και των διαπραγματεύσεων εκεί αποκινούμε ένα διορθωτικό το οποίο υιοθετήσαμε για το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής που γνωρίζουν τα σχετικά ισχυώδης. Όσοι είναι τώρα εδώ θα ήθελα να μπορέσετε να το δεχτείτε διότι το πρώτο θέμα για τον καπνό είναι το πιο σημαντικό. Δεν γνωρίζω αν θα συμφωνήσει ο κύριος Σμίτ, ε, θα συμφωνήσει ο Σμίτ με αυτή την μικρή αλλαγή. Και θα ήθελα να σας ζητήσω λοιπόν να εγκρίνετε την τελική θέση εξ ονόματος ε, δικού μου και όλων των σχεδόν εισηγητών επίσης για την πρότασή μας για τις ε, τροπολογίες όσον αφορά τα σκάφη αναψυχής και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μετά στο να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία στους τριμερείς διαλόγους με το Συμβούλιο. Είναι μία και μόνο ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ας διασφαλίσουμε τώρα ότι όλα λειτουργούν σωστά. Κάποιοι από τους κοιόδης θέλουν να σχολιάσουν κάτι. Όχι, εντάξει, περνάμε αμέσως στην ψήφιση. Άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία για τα σκάφη αυτά αναψυχής. Άρχεται η ψηφοφορία, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. 27 ψηφίζουν, 28 άλλος που θέλει να συμμετάσχει στην ψηφοφορία. Μπορούμε και αυτούς να τους προσθέσουμε και τη Σουζάνα. Άλλους, ο κύριος Μπόρισοφ παρίσταται, εντάξει. Λοιπόν, πέρας ψηφοφορίας τώρα. 29 υπέρ, 31 υπέρ, επειδή η κυρία Ρόιτοβα και οι συνάδελφοι υπερψήφισαν σας ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη στον εισηγητή και στην ομάδα σκιωδών εισηγητών για τις διαπραγματεύσεις. Πολύ καλά, λειτουργούν λοιπόν τα πράγματα σωστά. Και περνάμε στη συνέχεια τώρα στο κύριο θέμα για την ψηφοφορία μας από σήμερα, που είναι η γνωμοδότησή μας για μια νέα πρόταση για τον καπνό, για τις ρυθμίσεις ε, και όσον αφορά τις διατάξεις. Η κυρία Χάντσλικ είναι η συγγήτρια. Θέλετε να πείτε κάτι πρωτού ψηφίσουμε. Έχετε τον λόγο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Πολύ σύντομα πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι ήταν ένα πολύ δύσκολο χαρτοφυλάκιο να καλυφθεί. Ένα θέμα που έχει φορτιστεί ε, συναισθηματικά. Θέλω να ευχαριστήσω τους Κιώδης ε, και όλους σας για τη συνεργασία σας και για τις καλές σας προθέσεις να εξευρεθεί ένας συμβιβασμός. Προσπάθησα εγώ από πλευράς μου να επικεντρωθώ στα θέματα ασφάλειας, στην ασφάλεια και στην προστασία της υγείας των ε, καταναλωτών και σε σχέση με την Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτών και ε, αγοράς, εσωτερικής αγοράς, με χαρά μπορώ να δω την δυνατότητα να υπάρξουν συμβιβαστικές προτάσεις, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι επικοδομητικό. Θέλω και πάλι να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία σας. Σας ψηφίσουμε τώρα, Πρόεδρε, λοιπόν. Ευχαριστώ. Right, Ωραία, να ξεκινήσουμε λοιπόν. Και θα ήθελα να πω, θα ξέρουμε αν θα πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά από πλευρά των επίσημασεων των ε, ε, σχεδόν εισηγητών. Έχουμε τις ε, τροπολογίες για διαγραφή, υπέρ, κατά, απορρίφθηκαν. Μετά έχουμε κάποιες ταυτόσιμες τροπολογίες, στην 11 και τα λοιπά, υπέρ αυτών, κατά, εγκρίθηκε σαφώς. Η τροπολογία 119 υπέρ, κατά, απορρίφθηκε. Τροπολογία 120 Φαντεκάμπ υπέρ, κατά, απορρίφθηκε. Τροπολογία 12 εισηγήτριες υπέρ. Θα πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε τη 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την ομάδα μου εγώ. Πέρας ψηφοφορίας απορρίφθηκε με μία ψήφο διαφορά και ε, μία αποχή δηλαδή. Τροπολογία 13 της εισηγήτριας 121 υπέρ κατά εγκρίθηκε. Τροπολογία 122 υπέρ κατά να ελέγξουμε σε αυτή τη φάση ηλεκτρονικά να δούμε ποιοι είναι οι αριθμητικοί ε, συσχετισμοί 122 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκε αυτή η τροπολογία. 123 και 124 καταπίπτουν. 125 υπέρ. Θα πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά και πάλι για αυτήν. 125 άρχεται η ψηφοφορία. Κάποιοι δεν ψηφίζουν ίσως πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκε με μία ψήφο διαφορά. Λοιπόν, για τη διαγραφή κυρία Ρόιτοβα, έτσι. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ζητήσω να ζητήσετε από τον κύριο εκεί που παίρνει φωτογραφίες με το κινητό του τηλέφωνο να σταματήσει να βγάζει φωτογραφίες με το κινητό του. Εντάξει. Είναι ανοιχτή δημόσια συνεδρίαση, αλλά έχετε όμως δίκιο, θα ήταν σκόπιμο νομίζω να μην φωτογραφίζουν σε σχέση με την ψηφοφορία με τέτοιο τρόπο τα μέλη. Τροπολογία 126 υπέρ, κατά, απορρίφθηκε. 127 υπέρ, κατά, και αυτή απορρίφθηκε. 128 υπέρ, κατά, απορρίφθηκε. Τροπολογία 129 υπέρ κατά απορρίφθηκε. 131 υπέρ κατά απορρίφθηκε. 130 τροπολογία υπέρ κατά απορρίφθηκε 132 υπέρ κατά απορρίφθηκε 136 υπέρ κατά απορρίφθηκε τροπολογία 134 υπέρ κατά απορρίφθηκε Τοπολογία 133 και 135 υπέρ αυτών. Κατά. Νομίζω πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. 133-135 ηλεκτρονικά από κοινού. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκαν. 137 είναι γλωσσικού χαρακτήρα. 138 στάιλερ. Υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. Ε, ε, η 14 της εισηγήτριας υπέρ κατά εγκρίθηκε. 139 υπέρ. Καταπίπτει, ε, εντάξει, καταπίπτει. Συγγνώμη. 140 Φαντεκάμπ υπέρ κατά εγκρίθηκε. 141 με προφορική τροποποίηση υπέρ κατά εγκρίθηκε. 143 υπέρ κατά απορρίφθηκε 142 υπέρ κατά εγκρίθηκε 144 υπέρ κατά απορρίφθηκε 145 υπέρ κατά απορρίφθηκε 146 με προφορική τροποποίηση υπέρ πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά νομίζω άρχεται η ψηφοφορία. 146 άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίθηκε με μία ψήφο διαφορά. 147 υπέρ. Και πάλι πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την 147. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 149 καταπίπτη 148 υπέρ, κατά, απορρίφθηκε, είναι σαφές το αποτέλεσμα. Ωραία. Περνάμε στο άρθρο 3 τώρα. Συμβιβασμός 1 υπέρ, κατά, εγκρίθηκε, είναι σαφές. Περνάμε στον συμβιβασμό 2 υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. Περνάμε στην 173 της κυρίας Ράπτη, υπέρ. Εγκρίθηκε. 172 ως προσθήκη, υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. 174 υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. 177 υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. 176 και 175 καταπίπτουν. Ε, η συμβιβαστική τροπολογία 3. Υπέρ. Υπέρ της 3 συμβιβαστική. Εντάξει, θα ελέγξουμε το συμβιβασμό. Νομίζω εγκρίθηκε, αλλά θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά γι' αυτό. Πέρας ψηφοφορία και εγκρίθηκε 22 υπέρ 13 εναντίον. Περνάμε στον συμβιβασμό 4 υπέρ, υπέρ της 4 συμβαστική τροπολογίας. Κατά. Σαφές ότι εγκρίθηκε και περνάμε στην συμβαστική 5 υπέρ κατά σαφές ότι εγκρίθηκε συμβαστική 6 υπέρ κατά σαφώς εγκρίθηκε και πάμε μετά στην τροπολογία 275 της κυρίας Στάιλερ στην σελίδα 13 14 τουλάχιστον στο δικό μου κατάλογο υπέρ της 275 κατά Απορρίφθηκε η 275. Συμβιβασμό 7. Υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. Συμβιβασμό 8. Υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. Συμβιβασμό 9. Υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. Συμβιβαστική 10. Υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 11. Υπέρ κατά θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά με όλους αυτούς τους συμβασμούς πρέπει να ελέγχουμε καμιά φορά συμβασμός 11 άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά έχουμε 36 που συμμετέχουν στην ψηφοφορία 21 υπέρ 14 εναντίον έτσι λοιπόν περνάνε οι συμβιβασμοί τροπολογία 35 της εισηγήτριας υπέρ κατά εγκρίθηκε, είναι σαφές. Πάμε στην 369, κοράτσα μπιτ υπέρ, κατά, απορρίφθηκε. 370 υπέρ, κατά, απορρίφθηκε. 371 έγκστρομ υπέρ. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά λοιπόν. 371 άρχεται η ψηφοφορία έγκστρομ 371. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε η τροπολογία Έγκστρομ 19 ψήφι υπέρ 15 εναντίον. Η 372 Τώρα μπορούμε να ψηφίσουμε αυτήν. Η 372 λοιπόν υπέρ. Και πάλι θα ελέγξουμε την 372. Ψηφίζουμε άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκε με 19 υπέρ 16 εναντίον. 372. Οι 371 και 372 εγκρίθηκαν και οι δύο. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά. Σαφές ότι εγκρίθηκε. Τροπολογία 373 της κυρίας Στάιλερ. Υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 413 κόμι. Υπέρ. Και πάλι θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την 413 της κυρίας Κόμη. Άρχεται. Πέρας. Μπορούμε να ψηφίζουμε πιο γρήγορα. Παρακαλώ να πατάτε τα κουμπιά σας πιο γοργά. Πέρας ψηφοφορίας. <laughs> Εγκρίθηκε 18 υπέρ 15 εναντίον 3 αποχές. Εντάξει. Η 412 αποσ... καταπίπτει. 415 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίθηκε. Είναι σαφές. Η 416 Ρόιτοβα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 417 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 418 υπέρ και πάλι θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται, ψηφίζουμε την 418. Ψηφίζουν 37 μέλη. Η, η τροπολογία της κυρίας Κόμη λοιπόν, πέρας ψηφοφορίας. Και το αποτέλεσμα εγκρίθηκε. 419 της κυρίας Κόμη. Υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Και αυτή εγκρίθηκε με την ίδια πλειοψηφία. 420 της κυρίας Βερνιό. Υπέρ. Κατά. Σαφώς εγκρίθηκε. Μάλιστα. Να ελέγξουμε πολύ καλά. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 420. 37 συμμετέχουν, 36 ψηφίζουν. Πέρας ψηφοφορίας έχετε όλοι τις κάρτες σας στις συσκευές. Λοιπόν, 20 <clears throat> υπέρ 16 εναντίον μία αποχή εγκρίθηκε. Συμβασμός 13 υπέρ κατά εγκρίθηκε, είναι σαφές. Και περνάμε τώρα στην τροπολογία 351 και την 452 υπέρ αυτών κατά εγκρίθηκαν. 453 υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. Σαφές. 454 υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. 455. Όχι, δεν θα την ψηφίσουμε. Τεχνικού χαρακτήρα, αλλά πρέπει να ψηφίσουμε, λέει ο βοθός τον πρόεδρο. Ευχαριστώ. Σωστά λέει ο Πρόεδρο. Λοιπόν, για να αποσαφηνίσουμε αυτό το θέμα, τι συμβαίνει. Αυτές οι τροπολογίες ε, προηγούμενα είχαν εγκριθεί. Έχουμε τεχνικού χαρακτήρα τροπολογίες σε τμήματα ψηφίζουμε εδώ και χρόνια τώρα για αυτά τα θέματα. Λοιπόν, τι θα κάνουμε, περνάμε στο δεύτερο τμήμα. Όχι, το δεύτερο τμήμα όλο και όλο. Λοιπόν, το δεύτερο. Το δεύτερο τμήμα μόνο για τα πενταετή περίοδο, για αυτή τη ε, διατύπωση, πέντε χρόνια, υπέρ, κατά, σαφώς εγκρίνεται. Πέντε χρόνια εγκρίθηκε και το ίδιο και για την 458. Πρέπει και αυτό πάλι να ψηφιστεί στο δεύτερο τμήμα. Δεύτερο τμήμα για πέντε χρόνια, υπέρ, κατά. Πέντε χρόνια λοιπόν και πάλι εγκρίθηκαν. Δεν ψηφίζουμε τα άλλα, εντάξει, πολύ καλά. Η 469 λέτε Α, εντάξει. Ε, βρίσκεστε πολύ μπροστά. 469 υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. 470 υπέρ. Είναι πολύ στενό το αποτέλεσμα. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά για να ελέγξουμε. Πιο γρήγορα να ψηφίζετε παρακαλώ, να πατάτε πιο γρήγορα τα κουμπιά πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκε με 19 ψήφους υπέρ 16 εναντίον μια αποχή. 471 Βαντεκάμπ. Άρχεται η ψηφοφορία επ' αυτής. 471. Νομίζω η ίδια πλειοψηφία θα είναι αλλά καλό είναι να ελέγχουμε. Πέρας ψηφοφορίας Μάλιστα, ίδια πλειοψηφία. Όχι, όχι, απορρίφθηκε μάλιστα αυτή τη φορά. 16 υπέρ 19 εναντίον. Πολύ καλά. Απορρίφθηκε. 16 υπέρ 19 εναντίον μια αποχή. Απορρίφθηκε. Καλά κάναμε και ελέγξαμε, έτσι δεν είναι. 472 λοιπόν. 472 υπέρ. Κατά. Σαφώς εγκρίθηκε. 473 υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε, είναι σαφές. 53 καταπίπτει, 474 υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. 475 καταπίπτει, 54 και 476 υπέρ αυτών, κατά, εγκρίθηκαν. 477 υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. 478 καταπίπτει αυτή, 479 υπέρ, κατά, απορρίφθηκε. 53 Α, 55 διορθώνει ο πρόεδρο. Ζητώ συγγνώμη λέει ο πρόεδρο, 55 υπέρ. Να ελέγξουμε καλύτερα. 55. Άρχεται η ψηφοφορία. Νομίζω ότι είχε εγκριθεί. Αλλά θα αναμείνουμε να δούμε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Πράγματι εγκρίθηκε 20 ψήφοι υπέρ 15 εναντίον. Εγκρίθηκε. Τώρα, αιτιολογική σκέψη 4, τροπολογία 56 υπέρ, κατά. Απορρίφθηκε. 57 υπέρ, και πάλι θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 57. 57 άρχεται η ψηφοφορία. Εντάξει, πολύ καλά, πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε με ισοψηφία 18-18. Καλά κάναμε και ελέγξαμε πάλι. 58, Σαλβίνη, υπέρ. Κατά. Σαφώς εγκρίθηκε. 59, υπέρ. Κατά, εγκρίθηκε. 60 καταπίπτει. Τροπολογία 1 της εισηγήτριας, υπέρ κατά εγκρίθηκε τροπολογία 2 της συγκήτριας υπέρ κατά εγκρίθηκε τροπολογία 61 υπέρ κατά εγκρίθηκε 65 υπέρ κατά εγκρίθηκε 62 ως προσθήκη υπέρ κατά εγκρίθηκε 63 καταπίπτει και 64 καταπίπτει, 66 Στάιλερ υπέρ κατά απορρίφθηκε 67 υπέρ κατά εγκρίθηκε τοπολογία 3 καταπίπτει και 69 καταπίπτει και 68 καταπίπτει όχι διορθώνει τον πρόεδρο ο βοηθός όχι 68 η 66 απορρίφθηκε Πρέπει να ψηφίσουμε την 69, ελέγχουμε. Και την 69 επίσης, τροπολογία Σαλβίνη, είναι συμβατή ως προσθήκη. Ψηφίζουμε την 69 πρώτα, υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 68 τώρα, επίσης. Και αυτή συμβατή, εντάξει. Η 68 τώρα λοιπόν, ψηφίζουμε υπέρ, κατά. Εγκρίθηκε, είναι σαφές. Τροπολογία 70, Όμπερμαϊερ, υπέρ, κατά. Απορρίφθηκε τοπολογίες 4 της εισηγήτριας και άλλων υπέρ κατά εγκρίθηκε τροπολογία 76 που πάμε μετά συγγνώμη 76 έτσι σωστό τροπολογία 76 υπέρ κατά απορρίφθηκε 77 υπέρ κατά απορρίφθηκε 79 που είναι συμβατή έτσι υπέρ, κατά, απορρίφθηκε. Τροπολογία 78, υπέρ, υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. Τροπολογία 83, υπέρ, κατά, απορρίφθηκε. Τροπολογία 5, υπέρ. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 5, άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Νομίζω είχε εγκριθεί, αλλά θα δούμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε με μία ψήφο διαφορά 18 υπέρ 17 εναντίον. Εγκρίθηκε. Οι 82 τώρα, 85, 86, 81, 87 και 80 και όλες αυτές λοιπόν καταπίπτουν έτσι. Πολύ ωραία. Τροπολογία 88 τώρα υπέρ. Υπέρ κατά. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 89 είναι προστίκη, ευχαριστώ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 91 υπέρ, κατά εγκρίθηκε. 92 υπέρ, κατά απορρίφθηκε. Τροπολογία 95 υπέρ, κατά εγκρίθηκε. Έτσι λοιπόν η 93 καταπίπτει, η 6 και 94 καταπίπτουν. Πάμε στην 97 υπέρ κατά. Εγκρίθηκε η 97. 98 τώρα υπέρ κατά. Απορρίφθηκε. 99 υπέρ κατά. Εγκρίθηκε. 7 καταπίπτει 7. 8 και 100 υπέρ αυτών κατά. Εγκρίθηκαν μετά τροπολογίες 10 και τα λοιπά δεν θα ψηφιστούν, είναι τεχνικού χαρακτήρα. 9 και 101 τώρα, ναι σωστό, 9 και 101 υπέρ αυτών. Κατά εγκρίθηκαν αυτές οι δύο. Και πάμε τώρα στην 106 τροπολογία, σωστό, υπέρ. Κατά απόχες εγκρίθηκε. 107-108. Η 107 πρώτα υπέρ. Κατά απορρίφθηκε. Η 108 υπέρ. Κατά Απορρίφθηκε. 109 υπέρ. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 109 άρχεται. Απορρίφθηκε. 18-18 ισοψηφία απορρίφθηκε. 110 τροπολογία υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. 111 καταπίπτει. 112 υπέρ. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 112. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται, ψηφίζουμε την 112. Θα ψηφίσουν οι 37 που είναι, συμμετέχουν ή όχι. Πέρας ψηφοφορίας, εν πάση περιπτώσει. Και αποτέλεσμα απορρίφθηκε με δύο ψήφους διαφορά. 17 υπέρ 19 εναντίον. Τοπολογία 113. 113 υπέρ Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά τώρα για την 113. Πέρας ψηφοφορίας. Και εγκρίθηκε η 113. 18 ψήφοι υπέρ, 17 εναντίον με μία αποχή. Μάλιστα. Περνάμε στα παρατήματα. Τροπολογία 480. Έγκστρομ υπέρ. Σηκώστε τα χέρια όσοι είσαστε υπέρ. Οι φιλελεύθεροι ψηφίζουν όλοι. Ευχαριστώ. Κατά. Εγκρίθηκε, σαφέστατο. Η 481 καταπίπτει. Πολύ καλά. Περνάμε τώρα στην τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία, τελική ψηφοφορία στην τελική πρόταση. Τελική γνωμοδότηση. Έτσι. 37 κάρτες είναι στις συσκευές, 37 πρέπει να συμμετάσχουν, 36 ψηφίζουν, ένας λείπει, τι γίνεται. Ωραία. Κάποιος επιτέλους τα κατάφερε. Πολύ καλά. Εγκρίθηκε. 23 ψήφοι υπέρ και 14 εναντίον. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Χάνσλικ. Λοιπόν, θα διαβιβάσετε την άποψη της Επιτροπής στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε τώρα την ε, ψηφοφορία για την έκθεση της κυρίας mm. Μπέρα τις ψηφοφορίες που αφορούν τις εκθέσεις της κυρίας Μπέρα για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα πρώτα Κυρία Μπέρα, θέλετε να πείτε τίποτα? Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ήθελα απλώ ε, να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν σε διατύπωση του κειμένου αυτή και ειδικότερα τους σκιώδεις εισηγητές. Πρέπει να πω ότι είναι ένα κείμενο το οποίο είναι ιδιαίτερο τεχνικό και απαιτούσε ιδιαίτερη προσπάθεια. Είμαι πολύ ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα των εργασιών αυτών και σας ευχαριστώ. Μάλιστα, λέει ο Πρόεδρο. Α αρχίσουμε την ψηφοφορία για την ε, γνωμοδότηση αυτή. 14 τοπολογία υπέρ. Λοιπόν, για να είμαστε σαφείς, αρχίζουμε πρώτα με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και μετά θα πάμε στα in vitro διαγνωστικά. Λοιπόν, μιλάμε για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τροπολογία 14. Έχετε μπροστά σα το σωστό κατάλογο ψηφοφορίας. Ωραία. Είναι λίγο δύσκολε οι ψηφοφορίες ε, σήμερα. Κυρία Πρέντερ είναι έτοιμη. Ωραία. Όλοι έτοιμοι. Λοιπόν, Τροπολογία 14. Υπέρ. Λοιπόν, για να δούμε γιατί κάποιοι έφυγαν. Αρχίζει η ψηφοφορία για τη 14. 35 ψηφίζουν. 36 κάρτες τώρα. 36 κάρτες αλλά μόνο 34, 35 ε, ψήφισαν. Εγκρίνεται. 21-12. Λοιπόν, 94 τη κυρία Παρβάνοβα. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 95. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 96 τη εισηγήτριας. Υπέρ. Κατά. Υπέρ, υπέρ, συγγνώμη. Υπέρ. Τη 96. Υπέρ. Στο υπέρ είμαστε ακόμα. Τη εισηγήτριας. Κατά. Εγκρίνεται. 97. Κορία Ντεκάμπος όσο προσθήκη υπέρ κατά εγκρίνεται 16 και 98 υπέρ κατά εγκρίνεται 99 υπέρ κατά απορρίπτεται να ελέγξουμε εγκρίνεται διορθώνει ο πρόεδρος αλλά να το ελέγξουμε καλύτερα Μπορείτε να ψηφίσετε λίγο πιο γρήγορα, παρακαλώ. Τώρα μόνο 33, 34 άτομα ψήφισαν. Εγκρίνεται. 100. Υπέρ. Νομίζω ότι καλύτερα να την ελέγξουμε την 100. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Μάλλον εγώ είμαι ο μόνος που ψήφισε υπέρ. Τέλος πάντων. 17 αποσύρεται. 18. Προφορική τροπολογία της εισηγήτριας. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 20. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 101. Σφαμπ. Υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 102 προφορική τροπολογία υπέρ κατά εγκρίνεται. 103 έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την 103. Πέρας. Απορρίπτεται. 104 αποσύρεται, 105 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Σαφέστατα 106 υπέρ κατά εγκρίνεται. 107 υπέρ κατά εγκρίνεται. 21 αποσύρεται. 22 υπέρ κατά εγκρίνεται. 108 υπέρ κατά εγκρίνεται. 109 υπέρ κατά εγκρίνεται. 110 υπέρ κατά εγκρίνεται 23 υπέρ κατά εγκρίνεται 24 υπέρ κατά εγκρίνεται 25 υπέρ κατά εγκρίνεται 112 και 113 υπέρ κατά εγκρίνεται 114 προφορική τροπολογία υπέρ κατά εγκρίνεται 26 υπέρ κατά εγκρίνεται 27 υπέρ κατά εγκρίνεται 28 υπέρ κατά εγκρίνεται 29 υπέρ κατά εγκρίνεται 30 Τι ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 31. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 115. Υπέρ. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά να, να την ελέγξουμε ηλεκτρονικώς. Μιλάω για την 115. Πέρα της ψηφοφορίας, απορρίπτεται. 116 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 117 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 118 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 32 υπέρ κατά εγκρίνεται 33 υπέρ κατά Συγγνώμη, πάω πολύ γρήγορα. 33. Ψηφίζουμε 33. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 34. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 35. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 36. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 119. Υπέρ. Κατά εγκρίνεται 120 υπέρ ε, καταπίπτει 37 υπέρ κατά εγκρίνεται 38 υπέρ κατά εγκρίνεται 39 υπέρ κατά εγκρίνεται 121 υπέρ κατά εγκρίνεται 40 καταπίπτει 123 κατά τμήματα ψηφοφορία άρα πρώτο τμήμα Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 122 καταπίπτει. 124 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 125 υπέρ. Καλύτερα να την ελέγξουμε την 125. Πέρα τη ψηφοφορία 19-15 εγκρίνεται. 126 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 127 υπέρ. Κατά. Δεν κατάλαβα ποιος ψήφισε τι. Τα χέρια σας ήταν ε, πολύ δύσκολα να τα καταλάβει κανείς. Έναρξη λοιπόν ε, ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, πέρας. 22-13 εγκρίνεται. 128 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 129 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 130 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 41 και 131 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται επίσης 132. Προφορική τροπολογία της κυρίας Πιετικά είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 42-133 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 134 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 135 υπέρ. Κατά εγκρίνεται 136 υπέρ, κατά, εγκρίνεται 137 υπέρ, κατά, εγκρίνεται 138 υπέρ, κατά, εγκρίνεται 139, καταπίπτει 140 υπέρ. Καλύτερα να την ελέγξουμε. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 140. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 141 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 43 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 142 καταπίπτει. 143 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 144. 144 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 45 καταπίπτει λοιπόν. 145 υπέρ. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την 145. 145. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Άλλαξε γνώμη το ΕΛΚ. 146 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 147. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 46 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 47 υπέρ κατά εγκρίνεται 148 υπέρ κατά απορρίπτεται 149 υπέρ κατά απορρίπτεται 150 υπέρ κατά εγκρίνεται 151 υπέρ κατά εγκρίνεται 152 υπέρ κατά εγκρίνεται η 48 καταπίπτεια 49 υπέρ κατά εγκρίνεται. Η 154 τώρα, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 50, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 155, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 51, υπέρ, Κατά. Εγκρίνεται. 156 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται 157 και 158 υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται 52 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται 159 και 160 υπέρ. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για να, μην, ε, για να ασκήσετε και πάλι τα δάχτυλά σας. Πάλι άλλαξε γνώμη το ΕΛΚ. Μήπως μπορείτε να μου δείχνετε από την αρχή τι ψηφίζετε με, πιο σαφή τρόπο. 161 δεν την ψηφίζουμε. Και τώρα έχουμε όλες αυτές τις τροπολογίες που θα ψηφίσουμε μαζί υπέρ. Κατά εγκρίνονται. Και πάμε τώρα στην 61. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 162 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 163 αποσύρεται. 164 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 165 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 166 υπέρ. Προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Α, καλύτερα να μου το ξαναδείξετε τα χεράκια σας για την 166. Κατά. Εγκρίνεται. 167 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Άρθρο 53. Προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 168. Προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 169. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Λοιπόν, μπορούμε όλα αυτά να τα ψηφίσουμε μαζί όλες αυτές του Κορέα Αντικάμπος από την 170 171, 172, 173, 174 και 175. Και την 177. Μπορούμε να τις ψηφίσουμε όλες μαζί. Είναι όλες του Κορέα Αντικάμπος. Όχι την 175. Μέχρι την 175. Πολύ ωραία. Ψηφίζουμε. Υπέρ όλων αυτών των τροπολογιών. Κατά. Όλες αυτές συγκρίνονται. Πάμε τώρα την 177 υπέρ κατά εγκρίνεται 62 της εισηγήτριας υπέρ κατά εγκρίνεται 178 της εισηγήτριας υπέρ κατά εγκρίνονται 67 63 διορθώνει ο πρόεδρος υπέρ κατά εγκρίνεται 179 υπέρ κατά εγκρίνεται 64 υπέρ κατά εγκρίνεται. 181 προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 180 ως προσθήκη υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 182 πίπτη. 65 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 183 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 66 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 67 υπέρ. Α, καταπίπτει 67. Την ψηφίζουμε την 67 της εισηγήτριας. Αυτό ελέγχαμε τώρα. Λοιπόν, 67 της εισηγήτριας. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 68 της εισηγήτριας. Υπέρ. Ε, καλύτερα να ελέγξουμε ηλεκτρονικός. 68 της εισηγήτριας. Πέρας της ψηφοφορία. 20 20-16 εγκρίνεται. 69 της εισηγήτριας. Υπέρ. Ηλεκτρονικός καλύτερα. Την 69 της εισηγήτριας. Παρακαλώ λίγο πιο γρήγορα αν μπορείτε. Μόνο 34 θέλουν να ψηφίσουν τώρα. Τέλος. Απορρίπτεται. 17-18. Λοιπόν. 184 σφάμπ υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 70 της συγγήτριας υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 71 υπέρ. Κατά εγκρίνεται 72 υπέρ κατά εγκρίνεται 73 υπέρ κατά εγκρίνεται 185 καταπίπτει 74 λοιπόν υπέρ κατά εγκρίνεται 75 καταπίπτει α όχι δεν, την, δεν καταπίπτει την ψηφίζουμε, την ψηφίζουμε 75 λοιπόν υπέρ κατά εγκρίνεται 187 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 186 είναι συμβατή με την 187. Άρα την ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 188 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 76 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 189 προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 190 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 191 προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 192 υπέρ. Καλύτερα να την ψηφίσουμε ηλεκτρονικώς την 192 για να μην χαζεύουμε. Άντε, 35 άτομα θέλουμε. Μπαράβο. Εκατόν ενενήντα τρία. Εβδομήντα οχτώ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Εβδομήντα εννέα. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Εκατόν ενενήντα τέσσερα εγκρίνεται. 195 αποσύρθηκε, 80 υπέρ κατά εγκρίνεται. 196 υπέρ κατά εγκρίνεται. 197 υπέρ κατά εγκρίνεται. 198 υπέρ κατά εγκρίνεται. 199 υπέρ. Κατά. Γκρίνεται. 200 υπέρ. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Η κυρία Γκέπχαρτ είναι κατά και ο κύριος Φάμπιον υπέρ. Άλλαξαν τα πράγματα. Ωραία, είμαστε 35, πέρα της ψηφοφορίας. Α, εγκρίνεται. For once. Once he supported his amendment. Yes, yes, you support your own amendment this time. 201. 201. Έναρξη ηλεκτρονική ψηφοφορία για τη 201. Πέρας. Δύο άτομα έχουν βάλει τις κάρτες τους, αλλά δεν ψήφισαν. Τέλος πάντων απορρίπτεται, με μία αποχή. 202 τώρα. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Στην 81 πάμε τώρα και τη 203 υπέρ, κατά, εγκρίνονται. 201 και 82 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 82 καταπίπτει τελικά. 83 υπέρ, Κατά. Εγκρίνεται. 84 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 205 συμβατή υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 85 της εισηγήτριας υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 86 και 206 υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. 207 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 208 υπέρ κατά εγκρίνεται. 209 υπέρ κατά εγκρίνεται. Λοιπόν, 210 υπέρ κατά εγκρίνεται, 211 υπέρ κατά εγκρίνεται, 87 αποσύρεται, 212 υπέρ κατά Εγκρίνεται και τώρα πάμε σε αιτιολογικές σκέψεις. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 3 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 88 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται 4 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται 5 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται 6 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται 89 υπέρ. Κατά εγκρίνεται 7 υπέρ κατά εγκρίνεται 90 υπέρ κατά εγκρίνεται 91 υπέρ κατά εγκρίνεται 8 υπέρ κατά εγκρίνεται 9 υπέρ κατά εγκρίνεται 10 υπέρ κατά εγκρίνεται 11 υπέρ κατά εγκρίνεται 12 υπέρ κατά εγκρίνεται 92 υπέρ κατά εγκρίνεται 13 συμβατή υπέρ κατά εγκρίνεται 93 υπέρ κατά απορρίπτεται να ψηφίσουμε τώρα το σύνολο της γνωμοδότησης ε, ηλεκτρονικός 36 τώρα ψήφισαν. Μπράβο. Πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. 32 ψήφοι υπέρ. Καμία ψήφος κατά και 4 αποχές. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Μπέρα. Και τώρα προχωράμε.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 η δεύτερη έκθεση της κυρίας Μπέρε. Ξεκινάμε την τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 51 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 52 προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 53 υπέρ κατά εγκρίνεται 54 υπέρ κατά εγκρίνεται 55 υπέρ κατά εγκρίνεται 56 υπέρ κατά εγκρίνεται 57 υπέρ κατά εγκρίνεται 10 του εισηγητού υπέρ κατά εγκρίνεται 58 του κ. Φόξ υπέρ κατά απορρίπτεται 59 υπέρ κατά εγκρίνεται 11 είναι συμβατή υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά εγκρίνεται. Μπορούμε να τις βάλουμε μαζί κάποιες τροπολογίες. 12, 13, 14, 63, 15, 64, 65 και 67. 16 λέει ο πρόεδρος. Πώς σας φαίνεται αυτό όλες μαζί. Υπέρ κατά εγκρίνονται όλες 17 προφορική τροπολογία υπέρ κατά εγκρίνεται 18 υπέρ κατά εγκρίνεται 19 υπέρ κατά εγκρίνεται 20 υπέρ κατά εγκρίνεται 66 τροπολογία 66 υπέρ κατά απορρίπτεται 67 υπέρ, υπέρ, κατά, νομίζω, κατά, απορρίπτεται, απορρίπτεται. Τοπολογία 68 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τοπολογία 69 υπέρ, υπέρ, κατά, απορρίπτεται σαφώς. 70 υπέρ, κατά, απορρίπτεται 21 υπέρ κατά εγκρίνεται 22 υπέρ κατά εγκρίνεται 71 υπέρ κατά εγκρίνεται 72 υπέρ κατά εγκρίνεται εγκρίθηκε 58 όχι Ψηφίζουμε λοιπόν την 73. 73 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 75 υπέρ, κατά, ...75 υπέρ... ...κατά εγκρίνεται... ...23 που είναι συμβατή... ...θα ψηφίσουμε υπέρ... ...κατά εγκρίνεται... ...74 υπέρ... ...κατά εγκρίνεται... Πάμε να δούμε αν μπορούμε να βάλουμε κάποιες μαζί τροπολογίες. Όχι. Καλώς. 24. Υπέρ. Α, συγγνώμη, 76 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 77 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 78 υπέρ κατά εγκρίνεται ομαδικά κάποιες 26 να δούμε μέχρι θα φτάσουμε 26, 27 79 28, 29 80 μέχρι 80 καλώς 30 και 31 και 81 εντάξει ωραία ψηφίζουμε όλες μαζί λοιπόν υπέρ κατά Όλες εγκρίνονται. Ευχαριστώ πολύ. Στην 82 προφορική τροπολογία τώρα υπέρ. Κατά εγκρίνεται 83 προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά εγκρίνεται 84 υπέρ. Κατά εγκρίνεται 85 υπέρ. Κατά απορρίπτεται 86 υπέρ. Κατά απορρίπτεται 87 υπέρ κατά εγκρίνεται. Να πάρουμε όλες τις ε, τροπολογίες Κορέτα κάπως μαζί, 88, 89, 90, 91, 92 και 93 μαζί. Και 95 και 96, ωραία. Πάμε λοιπόν. Όλες αυτές λοιπόν από 88 μέχρι 96 υπέρ, κατά, όλες εγκρίνονται. 32 και 97 υπέρ, κατά, εγκρίνονται 99 υπέρ κατά εγκρίνεται 33 υπέρ κατά εγκρίνεται 98 υπέρ κατά εγκρίνεται 100 προφορική τροπολογία υπέρ κατά εγκρίνεται 101 καταπίπτει έχουμε τώρα με μάδα τροπολογιών του συγκητού μπορούμε όχι καλώς 34 υπέρ κατά εγκρίνεται 35 υπέρ κατά εγκρίνεται 36 υπέρ κατά εγκρίνεται 37 υπέρ κατά εγκρίνεται 38 υπέρ κατά δεκτή 39 υπέρ κατά δεκτή 40 υπέρ κατά δεκτή 102 υπέρ κατά δεκτή 41 ταυτόσημη ταυτόσιμη τροπολογίες με την 103 υπέρ κατά εγκρίνονται 42 υπέρ κατά εγκρίνεται 104 υπέρ κατά εγκρίνεται θέλουμε να τις πάρουμε μαζί αυτές όχι 43 υπέρ κατά εγκρίνεται 44 υπέρ κατά εγκρίνεται 45 υπέρ κατά εγκρίνεται 46 υπέρ κατά εγκρίνεται 105 κατά πίπτη συνεπώς 47 υπέρ μπλοκ μαζί 47 106 107 108 109 110 και 111 μαζί και 112 και 113 μέχρι τη λογική σκέψεις λοιπόν. Όλοι ικανοποιημένοι. Ωραία. Όλοι είναι υπέρ. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνονται όλες. Πάμε σε ιδεολογικέ σκέψεις λοιπόν. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 48 υπέρ κατά υπέρ ξανά 48 υπέρ κατά μισό λεπτό ας κάνουμε έλεγχο μπερδευτήκαμε τροπολογία 48 της κυρίας Βάισκερμπερ άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 15 υπέρ, 18 κατά. 49 μπορούμε να ψηφίσουμε τώρα υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 3 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Και 50 του κυρίου Μάντους. Άρχεται η ψηφοφορία για την 50. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Πέρας απορρίπτεται 18 υπέρ 18 κατά πολύ σκληρή μάχη ψηφίζουμε λοιπόν για την γνωμοδότηση στο σύνολό τη. άρχεται η ψηφοφορία Ποιος δεν ψήφισε, μόνο 34 ψήφισαν. 35 ανεβαίνουν οι αριθμοί πέρα ψηφοφορίας. 31 υπέρ. Καμία κατά και 4 αποχές. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Μπάρα. Σίγουρα θα εργαστείτε για να στήξετε θέση μας στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Μάντρος για την Επιτροπή Πολιτισμού για τα δικαιώματα που αφορούν συλλογικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο εισηγητής θέλει να πει κάτι. Να ξεκινήσουμε με την ψηφοφορία. Να ξεκινήσουμε και ευχαριστώ όλους διότι συμφωνήσαμε εφ' όλων. Ευχαριστώ. Right, let's go. Πρόεδρος, πολύ καλά. Ξεκινάμε. Τροπολογίες τροπολογίες 93 υπέρ κατά εγκρίθηκαν 95 υπέρ θα ψηφίσουμε την 95 Άρχεται η ψηφοφορία στην 95. Παρακαλώ πιο γρήγορα να ψηφίζουμε. Θα ήταν επικοδομητικό πιο γρήγορα. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε ισοψηφία 17 υπέρ 17 εναντίον. 96 Άρχεται η ψηφοφορία, ψηφίζουμε την 96. Παρακαλώ, πιο γρήγορα να πατάτε τα κουμπάκια. Παρακαλώ, συνεχίστε γρήγορα. 33 συμμετέχουν, 37 είμαστε που πρέπει να ψηφίσουν. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε με μία ψήφο διαφορά. 97 Φερχέιεν. Άρχεται η ψηφοφορία πάλι. Οι πλειοψηφίες μετακινούνται από ό,τι φαίνεται. Άρχεται η ψηφοφορία στην 97. 36 ψηφίζουν. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 18-18 ισοψηφία απορρίφθηκε. Δεν ξέρω. Κάποια κάρτα δεν συμμετέχει. Βρίσκεται στη συσκευή. Την ξέχασε κάποιος εκεί και δεν ψηφίζει. Ας το δει κάποιος. Εντάξει, συμβασμός 12 υπέρ κατά εγκρίθηκε. Τροπολογία 102 υπέρ κατά εγκρίθηκε. 103 υπέρ κατά απορρίφθηκε συμβιβασμός 14 υπέρ κατά εγκρίθηκε τροπολογία 106 υπέρ κατά απορρίφθηκε 13 εισηγητού υπέρ κατά εγκρίθηκε συμβιβασμός 44 υπέρ κατά εγκρίθηκε συμβιβασμός 15 υπέρ κατά εγκρίθηκε 110 Φερχάγιαν υπέρ κατά εγκρίθηκε συμβιβασμός 16 υπέρ κατά εγκρίθηκε πάμε στην τροπολογία 115 Ροσφόρ να μου πείτε εδώ τι θα πρέπει να γίνει. Άρχεται η ψηφοφορία, ψηφίζουμε την 115. Για να δούμε τι θα γίνει. Πέρας ψηφοφορίας συμμετέχουν 36. Απορρίφθηκε με δύο ψήφους διαφορά. Διαφορά 19 εναντίον 17 υπέρ. Απορρίφθηκε 116 υπέρ. Κατά. Και πάλι ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Είναι πολύ μικρές οι διαφορές. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 116. 36 συμμετέχουν. 35 τώρα συμμετείχαν, απορρίφθηκε. 17-17 ισοψηφία απορρίφθηκε. 117 βερνιό υπέρ κατά απορρίφθηκε, είναι σαφές. Συμβιβασμός 17 υπέρ κατά εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 18 υπέρ κατά εγκρίθηκε. 126 υπέρ υπέρ. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά και πάλι. Νομίζω εγκρίθηκε. Ψηφίζουμε την 126. Άρχεται η ψηφοφορία. 35 συμμετέχουν πέρας ψηφοφορίας τώρα. Εγκρίθηκε 21 ψήφοι υπέρ, 15 εναντίον, 127 υπέρ, κατά. Εγκρίθηκε με την ίδια πλειοψηφία, 128 Σάλτε Μόζε υπέρ, κατά. Εγκρίθηκε με την ίδια πλειοψηφία. 15 εισηγητού υπέρ κατά θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά ψηφίζουμε την 15 ηλεκτρονικά άρχεται 15 πέρας ψηφοφορίας αποτέλεσμα εγκρίθηκε 130 καταπίπτη η 129 έγκστρομ υπέρ κατά εγκρίθηκε Συμβασμός 19 υπέρ κατά εγκρίθηκε είναι σαφές 134 τροπολογία υπέρ κατά απορρίφθηκε 135 υπέρ κατά εγκρίθηκε συμβασμός 20 υπέρ κατά εγκρίθηκε 21 συμβασμός υπέρ κατά εγκρίθηκε 18 υπέρ κατά εγκρίθηκε 139 υπέρ κατά απορρίφθηκε 140 υπέρ κατά εγκρίθηκε 141 υπέρ κατά εγκρίθηκε 142 υπέρ καταπίπτει 142 ε. Μάλιστα. Περνάμε στο συμβασμό 23. συμβασμό 23 υπέρ. Υπέρ συμβασμό 23 κατά εγκρίθηκε 147 και 148 υπέρ αυτών κατά απορρίφθηκαν συμβιβασμός 24 υπέρ κατά εγκρίθηκε συμβιβασμός 25 υπέρ κατά εγκρίθηκε. Μια στιγμή. Συμβιβασμός 25 έτσι υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε μάλιστα. Συμβιβασμός 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 156 έγκστρομ υπέρ. Να ελέγξουμε όμως ηλεκτρονικά ψηφίζουμε την 156. Άρχεται. Νομίζω απορρίφθηκε. Θα δούμε. Πέρας ψηφοφορίας. 34 συμμετείχαν τώρα. Απορρίφθηκε με μία ψηφοδιαφορά. διαφορά. 157 υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε, είναι σαφές. 21 τροπολογία υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. 22 και 158 υπέρ αυτών. Και πάλι είσαστε υπέρ. Τι γίνεται. Κατά, ε. Ε, εντάξει. Θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 22 και 158 ηλεκτρονικά. Άρχεται. 22 και 158. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκαν με 17 ψήφους υπέρ και 17 κατά ισοψηφία. Η μία ψήφος ε, χάθηκε. 159 υπέρ κατά εγκρίθηκε. 160 υπέρ κατά εγκρίθηκε. Συμβασμός 27. Συμβασμός 27 υπέρ κατά εγκρίθηκε. Συμβασμός 28 υπέρ κατά εγκρίθηκε. Τροπολογία 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 164 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 165 αυτόματα εγκρίνεται έτσι. Ωραία, πάμε στην 25 τώρα. Τώρα 25, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 166 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 26, αποσύρθηκε αυτή. 167 υπέρ, κατά, απορρίφθηκε. Συμβασμός 29 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 170 τροπολογία υπέρ, όχι, όχι. Έχουμε ένα. Περνάμε στο συμβιβασμό. Συμβιβασμό 30 κατευθείαν. Συμβιβασμό 30 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 34 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 28 αποσύρθηκε. Πάμε στο συμβασμό 31 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Συμβασμός να ελέγξουμε. Εντάξει. Ψηφίζουμε το συμβιβασμό 31. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Με ισοψηφία 17-17 απορρίφθηκε. Ψηφίζουμε την 176 τροπολογία. 176 υπέρ. Θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 176 ηλεκτρονικά. Άρχεται. 176. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα εγκρίθηκε. 19 ψήφοι υπέρ, 16 εναντίον. Εγκρίθηκε. Ωραία. Συμβασμός 32 υπέρ. Κατά εγκρίθηκε. Η 141 είχε εγκριθεί. Ο συμβασμός 32 λοιπόν καταπίπτει ούτως ή άλλως πλήρως. Καταπίπτει. Επειδή διαγράφηκε η αντίστοιχη παράγραφος, έτσι σωστό, πρέπει να ψηφίσουμε τις επιμέρους τροπολογίες τώρα, μία-μία. 178, Έγκστρομ λοιπόν, υπέρ. Υπέρ της 178, κατά, απορρίφθηκε. 179, υπέρ, κατά, απορρίφθηκε. 181 υπέρ. Θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 181 ηλεκτρονικά. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας και αποτέλεσμα εγκρίθηκε με τρεις ψήφους διαφορά. Τι σημαίνει αυτό τώρα. Σημαίνει ότι Καταπίπτει 29 τροπολογία, έτσι. Αλλά η 180 είναι συμβατή. Εντάξει, ψηφίζουμε την 180 λοιπόν. 180 υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε η 180. Ωραία. Τροπολογία 30. 30 υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε η 30. Τροπολογία 182 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε 183 υπέρ κατά απορρίφθηκε 184 υπέρ Α, εντάξει, ωραία, δεν θα ψηφίσουμε την 184. Πάει αυτή. Συμβασμός 33 υπέρ κατά εγκρίθηκε. Πάμε στην τροπολογία 32 εισηγητού υπέρ κατά εγκρίθηκε. Καταπίπτει γιατί 34 υιοθετήθηκε, εγκρίθηκε. Ωραία. Λοιπόν, την 32 την εγκρίναμε πιο πριν. Σωστά. Πάμε στην 188. Όχι, καταπίπτει αυτή. Η τροπολογία 33 δεν, δεν υιοθετήθηκε. Ψηφίζουμε την 188 λοιπόν. Υπέρ υπέρ της 188 κατά εγκρίθηκε η 188 και η 189 είναι συμβατή και αυτή υπέρ της 189 κατά εγκρίθηκε ωραία περνάμε στην 190 τώρα υπέρ της 190 υπέρ κατά εγκρίθηκε 34 αποσύρθηκε 191 καταπίπτει συμβιβασμός 35 Πάμε στον συμβιβασμό 35 λοιπόν. Οι άλλες προηγούμενα κατέπεσαν υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίθηκε ο συμβιβασμός 35. Τροπολογία 37 υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίθηκε 38 υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίθηκε. Το ΕΚ ψήφισε για την 38, συμμετείχε. Εντάξει, ωραία, ευχαριστώ. Και πάμε τώρα, όλες οι άλλες καταπίπτουν αυτές που είναι στην Φεά στήλη. Α, ήταν για διαγραφή αυτή που λέτε. Εντάξει, ωραία. Τροπολογία 198 λοιπόν, υπέρ. Κατά εγκρίθηκε η 198. Και περνάμε, επειδή οι υπόλοιπε καταπίπτουν, πάμε στην συμβαστική τροπολογία 38 τώρα. Ωραία, υπέρ της 38. Κατά εγκρίθηκε αυτή. Πάμε στον συμβασμό 37 υπέρ. Κατά τα εγκρίθηκε. Πάμε στην τροπολογία 204. 44 διορθώνει ο πρόεδρος. Μάλιστα. 44, ναι. Σωστά. Τροπολογία 44, συμφωνείτε. Υπέρ, λοιπόν. Κατά. Εγκρίθηκε η 44. 210 καταπίπτει. 214 ε, τώρα. Υπέρ, κατά απορρίφθηκε 215 υπέρ κατά να ελέγξουμε ηλεκτρονικά ψηφίζουμε την 215 και άρχεται η ψηφοφορία ελέγχουμε έτσι οι πλειοψηφίε υπάρχουν πέρας ψηφοφορίες. εγκρίθηκε με τρεις ψηφούς διαφορά 19 υπέρ 16 εναντίον εγκρίθηκε 216 λοιπόν τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 217 υπέρ κατά απορρίφθηκε τροπολογία 45 εισηγητού υπέρ κατά εγκρίθηκε όλες οι άλλες καταπίπτουν πάμε στον συμβιβασμό 39 υπέρ κατά σαφώς εγκρίθηκε 223 υπέρ κατά εγκρίθηκε. Συμβιβασμό 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 230 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 231 υπέρ κατά Θα επαναλάβουμε. 230 συγγνώμη. 231 λέγεται στον πρόεδρο. Συγγνώμη. 231 λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφές και θα πρέπει να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την 231. Πέρας ψηφοφορίας. Και αποτέλεσμα απορρίφθηκε. 232 τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Όχι, εγκρίθηκε διορθώνει ο πρόεδρος. Εγκρίθηκε, μάλιστα. Συμβιβαστική τροπολογία 41 υπέρ. Συμβιβαστική τροπολογία 41 υπέρ. Μάλιστα. Συμβιβασμό 41 ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας και αποτέλεσμα εγκρίθηκε μάλιστα. Και έτσι πάμε στην 234 τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. 235 υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. 236 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 237 υπέρ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. Η 238 υπέρ κατά απορρίφθηκε. Η 51 εισηγητού υπέρ κατά απορρίφθηκε. Συμβιβασμό 42 υπέρ κατά εγκρίθηκε. 240 υπέρ κατά εγκρίθηκε. Συμβιβασμό 43 υπέρ κατά εγκρίθηκε. 54 υπέρ κατά εγκρίθηκε 55 υπέρ κατά εγκρίθηκε 242 αποσύρθηκε προφορική τροποποίηση τώρα Μάντερς και Μακλάκιν στο 41 υπέρ κατά εγκρίθηκε σαφώς Πάμε τώρα σε αιτιολογικές σκέψεις. Τροπολογία 56 υπέρ, κατά, συμβιβασμός 1 υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. Πάμε στη συνέχεια στον συμβιβασμό. Όχι, έτσι, ωραία. Πρέπει να πάμε στην 59 και 60 για διαγραφή. Τροπολογίες 59 και 60 υπέρ αυτών. Κατά εγκρίθηκαν. Πάμε στο συμβασμό 3 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε ο συμβασμός 3. 63 τροπολογία υπέρ. Κατά εγκρίθηκε. 64 κατά πίπτη. Τροπολογία 4. συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά εγκρίθηκε. 67 υπέρ κατά εγκρίθηκε. 68 υπέρ κατά απορρίφθηκε. 69 υπέρ κατά απορρίφθηκε. 70 υπέρ κατά εγκρίθηκε. 71 υπέρ κατά απορρίφθηκε. 3 υπέρ. Τι είπατε. Λοιπόν, 71. Ελέγχουμε και ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 71. Άρχεται. 71 λοιπόν. Ψηφίσατε όλοι. Ψηφίστε όλοι. 35 τώρα. Πρέπει να κλείσουμε την ψηφοφορία. Κλείνεται. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Η 3 καταπίπτει. Συμβασμός 5. Υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. Συμβασμός 6. Υπέρ. Κατά εγκρίθηκε. Τροπολογία 5 εισηγητού υπέρ κατά εγκρίθηκε. Συμβασμός 7 υπέρ κατά εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 8 υπέρ κατά εγκρίθηκε. Τροπολογία 6 υπέρ κατά εγκρίθηκε. 80 τι γίνεται, καταπίπτει αυτή. Η 7 εγκρίθηκε, έτσι, ευχαριστώ. Όχι, όχι, δεν εγκρίθηκε, λέγεται στον Πρόεδρο, αποσύρθηκε. Μάλιστα. Ψηφίζουμε τώρα την 80 υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε η 80. Συμβιβασμό 9 υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 81 υπέρ. Υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 9. Μια στιγμή. Μια στιγμή. Ωραία. Είχε ήδη υιοθετηθεί η 9. Η 82 καταπίπτει λοιπόν. Η 83 τώρα λοιπόν. 83 υπέρ κατά. Απορρίφθηκε. Συμβασμός 10 υπέρ κατά εγκρίθηκε. Τροπολογία 85 υπέρ κατά εγκρίθηκε. Συμβασμός 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 88 Τι έγινε με την άλλη, εγκρίθηκε 238 ή όχι. Να ελέγξουμε. Λέει εγκρίνεται αν έχει υιοθετηθεί, αν έχει εγκριθεί 238. Ας ψηφίσουμε ούτως ή άλλως. Είναι πιο εύκολο. Δεν είχε εγκριθεί 238. Λοιπόν, 88 ψηφίζουμε. Τροπολογία 88. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Σαφώς εγκρίθηκε. Θα ελέγξουμε διπλά τώρα, ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία, ψηφίζουμε την 88 εντάξει 88 37, 35, 34 συμμετέχουν πέρας ψηφοφορίας 18 υπέρ 4 εναντίον 12 αποχές μάλιστα εγκρίθηκε 89 τροπολογία είναι όμως γλωσσικής διατύπωσης θέμα μόνο 89 εν πάση περιπτώσει υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 91 υπέρ κατά απορρίφθηκε αυτή. Και τώρα ψηφίζουμε, να ελέγξουμε λέτε, 91, άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά, εντάξει. 91 ηλεκτρονικά. Λοιπόν, 91. Τροπολογία 91 γρήγορα παρακαλώ να ολοκληρώσουμε. 31 ψήφισαν μόνο. Πού είναι οι υπόλοιποι. Δεν, ξέρετε τι να ψηφίσετε. Εντάξει πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε λοιπόν. 31 όλοι και όλοι συμμετείχαν. Έχουν φύγει κάποιοι. Τέλος πάνω. εν πάση περιπτώσει, ε, ψηφίζουμε το, τελικό ψήφισμα τώρα σε τελική ψηφοφορία. Σχέδιο γνωμοδότησης του κυρίου Μάντας. Κάποιος άλλος θέλει να συμμετάσχει. 35 κάρτες έχουμε. 34. 35. Ποιος είναι εκείνος που βάζει βγάζει την κάρτα του στη συσκευή. Πέρας ψηφοφορίας. Κύριε Σμιτ. 34 υπέρ. Κανείς εναντίον. Μία αποχή. Συγχαρητήρια. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Μάντες. Πολύ καλά. Εξαιρετικά. Και προχωράμε στην τελική, στις τελευταίες ψηφοφορίες. Για την ψήφισμα για την ψηφιακή ενιαία αγορά, ο κύριος Αρίας και άλλοι την ετοίμασαν. Νομίζω ότι ο κόσμος ξέρει, μπορούμε να προχωρήσουμε γρήγορα ελπίζω και θα δούμε αν μπορούμε να βάλουμε ομαδικά κάποια, κάποιες ψηφοφορίες. Παράγραφος 1, τροπολογία 22 υπέρ, κατά εγκρίνεται.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 Are two voting lists on this. Right. I'm on version 4. Okay, all right. Uh, amendment 24. Τροπολογία 24 λοιπόν. Μάλλον 23. Α, 24 λοιπόν, υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 86, όσον εκρίθεται την Επιτροπή Απασχόλησης. Τροπολογία 25, υπέρ κατά εγκρίνεται 26 υπέρ κατά εγκρίνεται 27 υπέρ ας κάνουμε έναν έλεγχο τροπολογία 27 λοιπόν άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 18-15 Τροπολογία 28 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 81. 81 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 32 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. υποτιτλός υπέρ κατά εγκρίνεται συμβαστική 1 υπέρ κατά εγκρίνεται 94 δεν ψηφίζουμε συμβαστική 2 υπέρ κατά εγκρίνεται συμβαστική 3 υπέρ κατά εγκρίνεται τροπολογία 91 ρίπτεται 33 υπέρ κατά εγκρίνεται 95 ψηφίζουμε υπέρ κατά απορρίπτεται τροπολογία 34 υπέρ κατά εγκρίνεται τροπολογία 57 υπέρ κατά απορρίπτεται τροπολογία 58 υπέρ κατά εγκρίνεται τροπολογία 59 υπέρ κατά εγκρίνεται τροπολογία 60 και 61 μαζί υπέρ κατά εγκρίνονται η 60 και 61 35 υπέρ κατά εγκρίνεται 36 υπέρ κατά εγκρίνεται 37 υπέρ κατά εγκρίνεται 38 υπέρ κατά εγκρίνεται 62 39 υπέρ κατά εγκρίνεται 40 υπέρ κατά εγκρίνεται 51 θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά διότι είναι κρίσιμο θέμα αυτό για πολλούς Ξέρω το ιστορικό. Άρχεται η ψηφοφορία για την 51. 51. Ψηφίστε όλοι παρακαλώ. Έχουμε μια κάρτα παραπάνω κάπου. Πέρασες; Πέρας. Εγκρίνεται. 17-15 και δύο εποχές. Μικρή διαφορά. Το ίδιο για την 52. Άρχεται η ψηφοφορία για την 52. ...52. Ψηφίσατε όλοι. Μόνο 33-34. Ωραία πέρας. Γκρίνεται 29-3. 56 υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. 41 υπέρ υπέρ θα γίνει ηλεκτρονική ψηφοφορία στη 41 νομίζω πέρας εγκρίνεται 18-16 42 υπέρ κατά εγκρίνεται 49 73-75 αφήνουμε 74 υπέρ κατά εγκρίνεται 43 υπέρ κατά εγκρίνεται 44 υπέρ κατά 76 78 76-77-88 δεν ψηφίζονται 45 σε τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά εγκρίνεται δεύτερο τμήμα ψηφίζουμε ηλεκτρονικά το δεύτερο τμήμα ψηφίστε λίγο πιο γρήγορα δεν έχουν πολύ χρόνο. 34 τώρα. Απορρίπτεται. 16-18. 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 46 και 47 υπέρ κατά απορρίπτεται απορρίπτονται μάλλον 48 προφορική τροπολογία υπέρ κατά εγκρίνεται τίτλος υπέρ κατά εγκρίνεται 53-54 τα αφήνουμε 55 υπέρ κατά εγκρίνεται απορρίπτεται συγγνώμη τίτλος υπέρ του δέχεται του τίτλου 63, 64, 65 τα λαμβάνουμε υπόψη εγκρίνονται αυτομάτως 66 υπέρ κατά απορρίπτεται 67 λαμβάνεται υπόψη πάμε τη λογική σκέψη 11 υπέρ κατά εγκρίνεται 69 εγκρίνεται 12 υπέρ κατά εγκρίνεται 70 δεν ψηφίσετε 72 υπέρ κατά απορρίπτεται 13 υπέρ κατά εγκρίνεται 14 κατά τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ, κατά εγκρίνεται 68, αντιπόψη 71 υπέρ, κατά εγκρίνεται 16 υπέρ, 16 φιλελεύθερη κατά απορρίπτεται, 17 υπέρ, κατά εγκρίνεται, 19 υπέρ, κατά εγκρίνεται, 18 υπέρ, α, καταπίπτει 20 υπέρ κατά εγκρίνεται 21 υπέρ κατά εγκρίνεται λοιπόν λογική αναφορές μαζί ψηφίζουμε όλες μαζί ωραία όλες τις τηλεγικές αναφορές τροπολογίες 1 10 μαζί υπέρ κατά εγκρίνονται όλες ψηφίζουμε τώρα ορίστε μια και η τροπολογία 51 πέρασε. Είναι ένα πρόβλημα που έχουμε στη σχέση με την ομάδα μου. Η ομάδα μου θα ήθελε το σύνολο του κειμένου του ψηφίσματος να το υπερψηφίσει επειδή υπάρχουν πολλά και πολύ καλά θέματα σε αυτό το ψήφισμα. Όμως προτού περάσουμε στην τελική ψηφοφορία τώρα το, σε αυτό το ένα σημείο στην Ολομέλεια πρέπει να κάνουμε ξεχωριστή ψηφοφορία για αυτό το σημείο. Πρέπει να το ζητήσω εδώ ρητά και κατηγορηματικά, διότι προβλέπουν οι κανονισμοί ότι αν υπάρχει ομοφωνία, λέει στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή, δεν θα υπάρχουν τέτοιε ξεχωριστέ ψηφοφορίε. Επειδή θέλει η ομάδα μου να υπερψηφίσει το τελικό κείμενο, παρακαλώ τι άλλε ομάδε να δεχτούν στην Ολομέλεια να έχουμε ξεχωριστή ψηφοφορία για αυτό το σημείο. Okay. Καλώς η ομάδα μου, μιλώ για την ομάδα μου και η κυρία Μακλόκεν εδώ που είναι σκιώδης, θα σα υποστηρίξει για ξεχωριστή ψηφοφορία στην Ολομέλη. Ελπίζω και άλλες ομάδες να συμφωνούν. Επιπίας βάσεως λοιπόν. Με αυτό που εδώ σημειώνουμε ψηφίζουμε το ψήφισμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ομόφωνα εγκρίνεται. Ευχαριστώ πολύ όλους. Εκ μέρους του κυρίου Αρίας και του υποφαινομένου για τη στήριξή σας. Να σας πω, για όσους δεν ήσασταν εδώ νωρίτερα, ότι η διάσκεψη των Προέδρων συμφώνησε μια ειδική συζήτηση για τη νέα ψηφιακή αγορά την Πέμπτη το πρωί τη επόμενη Ολομέλεια. Ελπίζω όλοι σα να ζητήσετε χρόνο αγόρευση για να έχουμε καλή παρουσία στην Επιτροπή. Πέρα τη ψηφοφορία με 10 λεπτά καθυστέρηση Πάμε στο επόμενο σημείο. Ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα το πρωί. Right. Uh, um, παρακαλώ, όσοι αποχωρείτε, παρακαλώ με λίγη ησυχία, γιατί εμείς θα εξετάσουμε τώρα το σχέδιο γνωμοδότησης του κυρίου Έγγελ προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου για την πρόσβαση των προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων χωρών σε εσωτερική αγορά της Ένωσης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Πολύ σημαντική πρόταση και θα ήθελα να μας πει ορισμένα πράγματα ε, ο εισηγητής, ε, ο κύριος Έγγελ, είναι εδώ οι σκιώδεις συζητές, Βάιλερ, Κρόιτσμαν, Ρούλε, Μακλάρκιν, Κύριε Έγγελ, λοιπόν, σας δίνω το λόγο να παρουσιάσετε το σχέδιο γνωμοδότησής σας. Ευχαριστώ, Μάλκολμ. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για πρόταση κανονισμού, είναι ένα σημαντικό έγγραφο ε, δεν είχαμε και πολλά να κάνουμε και δύο πιθανότητες υπάρχουν, ε, όπως συμβαίνει συνήθως. Ε, ή μπαίνει κανείς ε, σε μία μακροχρόνια μάχη ισχύως μεταξύ των επιτροπών του Κοινοβουλίου και δεν καταφέρνει τίποτα ή, εν περιπτώσει, εκτιμάς αυτό το οποίο έχει έχουμε αποδεχθεί ότι μπορούμε να ε, κάνουμε. Τέλος πάντων, έχω ένα μεγάλο πρόβλημα με το κινητό μου σήμερα το πρωί. Τέλος πάντων, δύο στοιχεία. Πρώτον, το σχέδιο γνωμοδότησης που υπέβαλα αρκείται σε αυτό που ούτως ή άλλως αποφασίσαμε να κάνουμε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής ΣΥΜΚΟ και τα υπόλοιπα τα αφήνω στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Επομένω δεν είναι και πολλά αυτά που έχω να πω. Όπως θα διαπιστώσατε κι εσείς διαβάζοντας τη γνωμοδότηση αυτή, είναι κάποια διαδικαστικά σημεία και κάποια ε, στοιχεία τα οποία μπορεί ε, κατά τη γνώμη μου να ε, τα διατηρήσουμε και σε σχέση με τη δουλειά που κάνουμε για τις δημόσιες συμβάσεις. Ελπίζω να υπάρξει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των δύο δεν αποτελεί μυστικό και αυτό είναι το δεύτερο που θα ήθελα να πω ότι αυτή η πρόταση κανονισμού δεν είναι ε, αγαπητή σε όλους ε, σε κάποιες πολιτικές οικογένειες ε, κάποιες πολιτικές οικογένειες δεν την αγαπούν και σε ορισμένα τμήματα της, του Κοινοβουλίου η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου δεν είναι πολύ ικανοποιημένη και ε, ουσιαστικά πέρα από το περιεχόμενο ε, είναι κάτι το οποίο έχει ε, καθυστερήσει πάρα πολύ. Η τελευταία μελέτη ε, εκτίμησης επιπτώσεων ε, που ζητήσαμε εμείς για το κείμενο αυτό δεν είναι πολύ θετική. Λέει ουσιαστικά ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν τίποτε να κερδίσουν από την έγκριση του κειμένου αυτού και επίσης ε, λέει και αυτό το ξέραμε και από πριν, ότι μπορεί να υπάρξουν και αντίπεινα από ε, άλλους ε, εταίρους που δεν συμφωνούν με αυτά που αναφέρονται. Εγώ πιστεύω στην αμοιβαιότητα και πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε να είμαστε βασιλικότεροι του βασιλέως. Ε, πρέπει να προσπαθούμε να ε, βρούμε τους φίλους μας σε όλο τον κόσμο. Εφόσον ε, έχουμε ανοίξει εμείς πολλές πόρτες, θα περιμέναμε και εκείνοι να κάνουν το ίδιο και δεν ξέρω αν ε, δεν μπορούμε να το πετύχουμε αυτό με διαπραγματεύσεις, δεν ξέρω αν μπορούμε πράγματι να, το πετύχουμε ε, με ένα τέτοιο κείμενο. Γιατί η μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων ε, δεν δείχνει κάτι τέτοιο ως πιθανό αποτέλεσμα. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για το κείμενο αυτό στο σύνολό του, μόνο για την πτυχή που μας αφορά ως Επιτροπή. Μέχρι τις 7 Ιουλίου έχετε νομίζω αρκετό χρόνο να μου πείτε την άποψή σας. Ε, εγώ επέλεξα να παραμείνω στο πλαίσιο της εντολής που έχουμε λάβει εμείς ως ε, Επιτροπή για να μην δημιουργήσουμε προβλήματα όταν θα πάει η γνωμοδότησή μας στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου και μετά μπορεί να έχουμε προβλήματα ε, αποδοχής της γνωμοδότησής μας. Τώρα, κατά πόσο οι συνάδελφοι συμφωνούν ε, ή όχι, εγώ θα έλεγα ότι θα ήταν καλό να συμφωνήσουμε, να διατηρήσουμε τα πράγματα όπως σας τα λέω, γιατί ε, αν παραμείνουμε στην εντολή που ε, έχουμε, θα κάνουμε τη δική μας ζωή ευκολότερη για να καταλήξουμε στο τελικό κείμενο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την σαφέστατη θέση σου ως προς αυτό. Συμφωνώ. Πρέπει να λύσουμε τα θέματα του άρθρου 50. Ε, έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε, όπως είπες και εσύ. Ας προχωρήσουμε τώρα με τους σκιώδεις εισηγητές. Ε, πρώτα η κυρία Βάιλερ. Ναι, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Έγγελ, έχω πράγματι σέβομαι το ότι περιορίζεστε στα θέματα του, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς. Δεν πρέπει να συζητήσουμε επί παντός του επιστητού και να τα συμπεριλάβουμε στην έκθεσή μας. Από πλευράς αρχής έχει απόλυτο δίκιο αυτή η θέση. Όμως η κατάσταση δεν είναι και τόσο σαφής όπως το προανέφερε ο Πρόεδρος. Διότι, καταρχήν, η ομάδα μου ναι μεν ήταν πάντα υπέρ του ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στοχεύει προς την ορθή κατεύθυνση, παρότι υπάρχουν πολλαπλά επικρίσεις, ιδιαίτερα από την γερμανική και ευρωπαϊκή οικονομία, ως κύκλους. Παρόλα αυτά είναι δύσκολο θεωρώ αυτή τη στιγμή να συνεχίσουμε έτσι στο μέλλον. Αν τη μελέτη επιπτώσεων του Κοινοβουλίου την δει κανείς από πιο κοντά. Τυχαία εχθές, όχι τυχαία, αλλά χθε ήμουνα στην Επιτροπή Εμπορίου και παρόλα αυτά από τον κύριο εισηγητή εκεί τι αναφέρθηκε. Πολύ έντονα αναφέρθηκε η μελέτη επιπτώσεων του Ευρωκοινοβουλίου που βρίσκεται σε μεγάλη αντίθεση με τη μελέτη επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι επιφυλάξεις και διαφωνίες και διαφορές μεταξύ των δύο μελετών αυτών, μελετών επιπτώσεων δεν άρθηκαν, δεν ε, ανταποδείχθηκαν στη συνεδρίαση αυτή της Επιτροπής Εμπορίου εξακολουθούν και υφίστανται αυτά τα προβλήματα τόσο έντονα ώστε η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή ή ο εισηγητής της συνέστησε σοβαρά προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το σύνολο αυτής της πρότασης να, να την αποσύρει, να αποσύρει το σύνολο αυτής της πρότασης. Και γι' αυτό και δεν το βρήκα παράλογο, ας το πω έτσι, δεν το βρήκα ασύνεπες, γιατί θα θέλαμε να έχουμε μια σοβαρή πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ευσταθή πρόταση με πολιτικά κριτήρια, κοινωνικά κριτήρια και παρόμοια κριτήρια, αν όμω δεν υπάρχουν τέτοιε προτάσει, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα σχετικό. Παρ' όλα αυτά όμω πρέπει, προτού σοβαρά συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση, πρέπει με τον κύριο εισηγητή επί της ουσίας να συζητήσουμε. Αν δηλαδή αυτή η στρατηγική θα τύχει συνέχεια να αποσυρθεί αυτή η πρόταση, επειδή ακριβώς ε, η υπόθεση ότι μέσω της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, δημιουργούνται λέει πολλές θέσεις, νέες θέσεις απασχόλησης και ιδιαίτερα από μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε αναδιόμενες χώρες και αυτή η προϋπόθεση δεν είναι πλέον δεδομένη, δεν ευσταθεί πλέον και αν αυτή η προϋπόθεση επί της οποίας οικοδομούμε και θεμελιωνόμαστε σε αυτήν δεν είναι δεδομένη, τότε πραγματικά το θεωρώ, πώς να το πω, το θεωρώ περιττό εκ του περισσού και αμφισβητήσιμο κιόλας να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με τέτοια υπόθεση εργασίας ως δεδομένο. Πρέπει να αποσαφηνίσουμε τι γίνεται. Από όλες τις πλευρές τονίστηκε αυτό χθες, ότι δηλαδή η νέα μελέτη επιπτώσεων του Ευρωκοινοβουλίου με πολύ, βασίζεται σε πολύ σοβαρά δεδομένα και μελέτες. Δεν είναι κάτι που ελαφρά την καρδία μπορούμε να απορρίψουμε και να πούμε δεν μας ενδιαφέρει. Πρέπει να μας ενδιαφέρει. Και γι' αυτό το λόγο επανέρχομαι κιόλας στα θέματα της πρώτης συζήτησης που θα θυμόσαστε ότι τότε είχα προτείνει ότι και είχα πει ότι ο σημαντικότερός μας εταίρος εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΠΑ δηλαδή, έχουμε το FTA που την επενούμε πολύ αυτή την συμφωνία εμπορίου τουλάχιστον αυτό να συμπεριληφθεί ώστε να έχουν ευκολότερα πρόσβαση οι ευρωπαϊκές εταιρείες στην ε, αμερικανική αγορά εργασίας. Τώρα τι γίνεται, δεν χρειαζόμαστε κάτι τέτοιο. Συμπέρασμα λοιπόν, πρέπει να αποσαφηνίσουμε ποια συνέχεια θα δώσουμε με την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή επ' αυτού του θέματος και μετά να αποφασίσουμε αν θα συμφωνήσουμε και ακολουθήσουμε την πρόταση ή όχι. Yes. Well, I'm... Uh, thank you. Thank you. Ευχαριστώ που μας ενημερώσατε όσον αφορά αυτά που συμβαίνουν στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Είναι σημαντικό και ίσως θα μπορούσε ο εισηγητής να σχολιάσει το εξελισσόμενο σενάριο. Άκουσα και εγώ τα ίδια, είχα ίδια εντύπωση από τον εισηγητή στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Είναι καλό που συζητήθηκε η έκθεση επιπτώσεων του Κοινοβουλίου. Θα σχολιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την οποία καλωσορίζω και ζητώ συγγνώμη δεν είχα χαιρετήσει τον ε, εκπρόσωπο της DG Mark. Δεν ξέρω αν από τη DG Trade αν ήρθε κάποιος. Θα αργήσουν να αργήσουν κι άλλο. Όπως καθυστερεί και η πρόταση άλλωστε. Καλώς. Ο κ. Κρόιτσμαν είναι επόμενος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Έγκελ για τη δουλειά που κάνατε σαν εισηγητής για το επίμαχο θέμα. Ο κ. Λέγκεγκάρντε μπορούσε να παρίσταται και συμφώνησε να παρουσιάσει την άποψή του. Λοιπόν, στην πρώτη εντάλλαξη απόψεων ο κ. Δίνκεγκάρτ κατέστησε σαφέ ότι πιστεύει ότι εξαίρεση ε, εξαιρέσει αυτού την αγορά τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω δεν θα οδηγήσει άνοιγμα τρίτων χωρών. Αντιθέτω, η χρήση του άρθρου 6 θα οδηγήσει σε αντίπεινα από τρίτε χώρε και θα θέσει διοικητικό άχθο επί των τοπικών αρχών. Γι' αυτό ο κ. Λίγκεγκάρτ προτείνει να διαγράψουμε το άρθρο 6 και να κρατήσουμε τη διαδικασία διαβούλευση που αναφέρεται στο άρθρο 8 8-10 όχι μόνο για να εξασφαλίσουμε ότι δεν κινδυνεύουμε από κατακαιρματισμό της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ενώσης, να εξασφαλίσουμε επίσης ότι δεν κινδυνεύουμε να έχουμε δύο αλληλοκαλυπτόμενες διαδικασίες. Οι Κινέζοι, παραδείγματος χάρη, μπορεί να, μπορεί να γίνει δεχτή μια θέση στο Λονδίνο και κινέζικη ε, προσφορά και στην Πράγα ή στο Λονδίνο να απορριφθεί κάπου και αλλού να, μην, ε, να γίνεται δεχτή και αλλού να απορρίπτεται. Οπότε το άρθρο 6 ε, έπρεπε να αλλάξει και να ελεγχθεί στο σχέδιο εκθέσεως. Κυρίως γιατί το άρθρο 6 είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ο εισηγητής ο κ. Κασπάρη δήλωσε σαφώς ότι πιστεύει ότι αλλαγή το άρθρο 6 ε, θα ανήκει στην Επιτροπή ΕΚΟ και θα έχουμε τεράστια ευθύνη αν θέλουμε να αλλάξουμε αυτό το κομμάτι του νομοθεσίας. Στο άρθρο 6 στην ΑΦΕΤ συζητήσαμε τον Μάρτιο το θέμα. Άλλο σημαντικό άρθρο που δεν συζητήθηκε. Ήταν το 7. Δυνατότητα τοπικής αυτοδίκησης να εξετάσει τι γίνεται με τις πολύ χαμηλές προσφορές. Ευχαριστούμε τον κύριο Άγγελ για αυτό το άρθρο. Είναι σημαντικότατη επιλογή που δίνουμε στην τοπική αυτοδίκηση. Σίγουρα συμπληρωματικέ πληροφορίε πρέπει να δίνονται από αυτόν που κάνει την προσφορά εάν είναι πολύ χαμηλή προσφορά. Ο κύριος Λέγκριντ πιστεύει ότι θα πρέπει να είναι υποχρέωση και όχι επιλογή όσον αφορά το να δίνει αυτός που κάνει την προσφορά και άλλες πληροφορίες. Αν δώσει, εάν οι πληροφορίες είναι ανεπαρκείς, πρέπει να για να εξηγήσουν την πολύ χαμηλή τιμή η τοπική αυτοδίκηση δεν πρέπει να έχει την επιλογή μόνο, αλλά πρέπει να είναι υποχρεωμένη να επανεξετάσει την προσφορά. Άλλα σημαντικά σημεία συζητήθηκαν. Αυτά που ανέφερα είναι κάποια σημαντικά σημεία που θέλει η Άλντε να αλλάχθουν στην επόμενη διαδικασία. Τέλος, εξού σημαντικό. Καλύτερο θα ήταν να μην έχουμε συγκανασμό τη της Ευρωπαϊκής αντί να έχουμε αδύναμη νομοθεσία. Πολλά κράτη-μέλη ήδη έχουν τέτοιες επιλογές στη δική νομοθεσία για να μπορούν να επανελέγχουν ανώμαλα χαμηλές φορές. Εάν θετήσουμε χαμηλότερο επίπεδο νομοθεσία, ίσως αποδυναμώσουμε κάποια νομοθεσία κρατών μελών. Διότι εδώ η κοινοτική νομοθεσία υπερέχει της εθνικής. Θα προτιμούσαμε λοιπόν καμία λύση καθόλου παρά κακή λύση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Πριν καλέσω την κυρία Ρούλε, να καλωσορίσω τον Άντερ Γέρτσεν από τη DG Trade. Έχουμε όλη την ομάδα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Ρούλε. Κύριε Κρόσμαν, με απογοητεύσατε πολύ. Είχα την ελπίδα ότι ο κύριο Λόκεγκαρτ και εσεί θα παραμένατε στην άποψή σας την πρόταση αυτή να την επαναπέμψουμε πίσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είχα καταλάβει στο παρελθόν από τον κύριο Λόκεγκαρτ. Και λυπούμε, θλίβομαι. Ε, τότε εντάξει, να περιμένουμε να δούμε θα με λυπούσε αν είχε αλλάξει την άποψή του. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι όχι μόνο η μελέτη επιπτώσεων του Ευρωκοινοβουλίου είναι υπέρ αυτού, αλλά αν δει κανεί τι αντιφάσει στη μελέτη τη Επιτροπή, τότε πρέπει να είμαστε υπέρ του ότι αυτή η πρόταση δεν είναι καλά διατυπωμένη. Δεν έχει εκπονηθεί καλά. Πέρα από αυτό πιστεύω ότι θέλω να αναφέρω κιόλα και τον εισηγητή. Το ότι δηλαδή εδώ τα προβλήματα στις διαπραγματεύσεις για το εμπόριο, για το διεθνές εμπόριο, θα πρέπει εκεί να επιλύονται τα προβλήματα και όχι εδώ σε πρώτη γραμμή να έχουμε ε, την, ε, τον επιμερισμό αυτού του έργου. Όχι μόνο δεν ωφελεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά είναι και επιπρόσθετο γραφειοκρατικό βάρος, επιπρόσθετη επιβάρυνση για τις ε, προμήθειες και τις ε, συμβάσεις αυτές. Γι' αυτό θα το υποστηρίζαμε αν πλειοψηφικά στο Κοινοβούλιο καταλήγαμε σε μια απόφαση να συστήσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσύρει αυτή την πρότασή τη. Παρ' όλα αυτά θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή, διότι επικεντρώθηκε στα ουσιοδέστερα θέματα ω ζητήματα σε σχέση με την Κοινοβουλευτική μα Επιτροπή. Δεδομένη της κατάσταση δεν απομένει τίποτα άλλο. Τι να κάνει δηλαδή ένα εισηγητή όταν η κατάσταση έχει ούτω. Ευχαριστώ λοιπόν τον εισηγητή. Θα θέσουμε το αίτημα για την επαναπομπή. Θα υπάρξει αυτό το αίτημα αλλά όταν θα, έχουμε στις θα έρθουμε σε επιμέρους τροπολογίες δεν είναι επίμαχα τα θέματα, παραμένουμε και έχουμε συμφωνία από αυτών. Ελπίζω ότι η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή θα αποφασίσει διαφορετικά λοιπόν. Ευχαριστώ. Ε, thank you. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μακλάρκεν. Όπως είπε και η συγγητής, είχαμε περιορισμένο πεδίο θεμάτων στην Επιτροπή. Είμαι σκιώδης του ECR στην Ίντα για το θέμα. Παρακολουθώ στενά από την αρχή το θέμα. Και πρέπει να τεθεί τέρμα σύντομα, ελπίζω. Διότι όπως δείχνει και η αξιολόγηση συνεπιών που ενισχύει και τις αρνητικές ε, μελέτες, ε, τα αρνητικά πορίσματα, λέει ότι δεν υπάρχει κάποια βάση για το προτινόμενο αυτό εργαλείο που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και θα είναι επιζήμιο περισσότερο ή την αγορά φοβάμαι και για τις επιχειρήσεις και έχω ανησυχίες για κάποιες ε, τροπολογίες για το σχέδιο γνωμοδότησης θα οδηγήσουν στην αύξηση της γραφειοκρατίας στη διαδικασία. Εν γέννη, πιστεύω ότι θα είναι κάτι κακό για τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και για την ανταγωνιστικότητα στην ενιαία αγορά. Μακροπρόθεσμος αντίκτυπος της πρότασης αυτής οδηγήσει σε αντίπεινα, κάτι πολύ επιζήμιο και θα πρέπει στην Επιτροπή αυτή να συζητήσουμε σοβαρά τον δεχόμενο απόρριψη και επαναπομπή τη πρόταση για περαιτέρω ανάλυση στην Επιτροπή ΙΝΤΕ. Και πιστεύω ότι το συμπέρασμα θα είναι γιατί εργαζόμαστε, επεξεργαζόμαστε κάτι το οποίο δεν έχει βάση ούτε είναι υποφελέ. Εν κατακλείδη περί αυτού πρόκειται, αλλά θέλω να ακούσω και το τι έχει να πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από αυτό. Καλώ. Άλλοι βουλευτέ θέλουν να συζητήσουν, να εκφράσουν άποψη. Ο κύριος Μπαλταζάρη. Κύριε Μπαλτασάρη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ βεβαίως τον Φρανκ Έγκελ για το σχέδιο γνωμοδότησης για μια πρόταση κανονισμού που θα έπρεπε να είναι κάτι σημαντικότατο για την οικονομική ανάκαμψη και την απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαφορά όμως και η συμμετρία που υπάρχει μεταξύ της πρόσβασης στην αγορά όσον αφορά τις δημόσιες προμήθειες της, της Ευρωπαϊκής Ένωσης 350 δις ευρώ και το κλείσιμα, το κλείσιμα που έχουν οι άλλες χώρες όσον αφορά τις προμήθειες είναι κάτι απτό. Δεν χρειάζονται αξιολογίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να καταλάβουμε ότι εμείς προσφέρουμε δυνατότητες ύψους 350 δις, στη ΣΥΠΑ για 170, στην Ιαπωνία 27 δις, η Κίνα είναι κλειστή αγορά για τους Ευρωπαίους. Γιατί αν διαβάσατε τους όρους αναγκαίους για μια ευρωπαϊκή επιχείρηση να μπορεί να πάει να εργαστεί στην Κίνα, στον τομέα στον οποίο είμαστε ισχυρότεροι, δηλαδή κατασκευές, οικοδομίες και σιδηρόδρομοι, είναι ουσιαστικά κλειστή αγορά. Και όχι μόνο, όπως έλεγε, και όπως φέτη στην εισήγησή σου, η οικονομική κρίση οδήγησε σε άλλε χώρε να θετήσουν μέτρα τα οποία είναι άκρως προστατευτικά, όπω Βραζιλία, Ρωσία, όπου το σωστά των προϊόντων. Ε, είναι πολύ δύσκολο να συμμετάσχουμε. Λοιπόν, αυτό είναι το πλαίσιο. Και η πρόταση θέλει να ενισχύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση στις διαπραγματεύσεις. Αλλά το γραφειοκρατικό άχθος που δημιουργούμε και αυξάνουμε το άχθος θεσπίζοντας αυτή την νομοθεσία. Αυτές οι ανησυχίε δεν είναι κάτι ίσονο σημασία. Όπως και οι μελέτες συνεπιών. Είναι πολιτικό και οικονομικό το πρόβλημα. Μετά, δεν κρύβομαι. Όπως γνωρίζουμε όλοι, ως συνήθω στο Συμβούλιο υπάρχουν κάποιες χώρες που φυσικά στηρίζουν τα δικά του συμφέροντα και προσπαθούν να εμποδίσουν να θετήσουμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση μια συνολική τοποθέτηση που θα είναι πολύ πιο παραγωγικό σαν τοποθέτηση και θα τονώνει καλύτερα την οικονομία και θα δημιουργεί θέσει απασχόλησης. Το θέμα της ανεργίας φαίνεται να μην έγινε πρόβλημα μόνο κάποιων χωρών, αλλά γενικό πρόβλημα. Πιστεύω λοιπόν και είμαι συγγητής εγμοδότης στην Επιτροπή, νομική, Επιτροπή Νομική, αλλά και στη δική μας Επιτροπή, στην ΙΜΚΟ, θα πρέπει να κάνουμε κάτι να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα. Τις ανησυχίες του εισηγητή Έγγελ τις ημερίζομαι ότι πράγματι σαν Επιτροπή δεν μπορούμε να παρεύουμε πολύ σε το κείμενο, όμως νομίζω ότι, πώς να το πω, θα μπορούσαμε να εισάγουμε κάποιες τροπολογίες ή διορθώσεις για να έχουμε μια πιο ισχυρή πολιτική θέση, κυρίως όσον αφορά το άρθρο 6 Εκεί ίσως κάπως πιο περιοριστική διάταξη θα μπορούσε να εισαχθεί. Εμείς στη Νομική Επιτροπή έχουμε εισαγαγεί εδώ δύο στοιχεία καινούρια ρυθμίζοντας τους, τις και τους διαγωνισμούς και σε περιπτώσεις όπου είναι, αφορούν ποσά κάτω 5 εκατομμύρια ευρώ. Για συμβάσεις κάτω των 5 εκατομμύριων ευρώ οι αναθέτους αρχές μπορούν να αποκλείσουν προσφορές από τίτλες χώρες αν είναι πάνω από 50 κάτω από 50 και να δούμε αν ε, μπορούν να υπάρχουν δυνατότητες αποκλεισμού. Αλλά και στις πολύ χαμηλές προσφορές, ανώμαλα χαμηλές, θεωρήσαμε και πιστεύουμε ότι ισχύει ότι πρέπει να δώσουμε πιο ε, στενή περιοριστική ερμηνεία στην προτινόμενη νομοθεσία. Θα πρέπει πάντα να δίνονται γραπτός πληροφορίες στους άλλους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό όταν θεωρεί η δίκηση ότι μια προσφορά είναι ανώμαλα χαμηλή. Χωρίς να επιστέψουμε επί των αναφερθέντων επιχειρημάτων, πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να στείλει ένα πολιτικό μήνυμα σαφές και για το εσωτερικό και για το εξωτερικό της Ένωσης. Για να ξεπεραστούν και οι συνηθισμένες αντιστάσεις των εθνικών συμφερόντων και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει διαπραγματευτικά εργαλεία πιο ισχυρά που θα επιτρέψουν να υπάρχει δυνατότητα να πηγαίνουμε στο τραπέζι των επαγματεύσεων για τους διαγωνισμούς όχι σε μειονεκτική θέση όπως είναι σημερινή. Δείχνουμε αν έχουμε μια αγορά ελεύθερη, εντελώς ελεύθερη. Δεν θέλουμε να εφαρμόσουμε μέτρα προστατευτικά, θα ήταν σφάλμα, αλλά πώς να αντιταχθούμε σε κάποιους που δεν άνοιξαν ποτέ την αγορά τους ή ε, υιοθέτησαν και μέτρα πρόσφατα για να κλείσουν περισσότερο τις αγορές τους. Νομίζω ότι είναι δύσκολο να φανταστούμε την απειλή ε, ε, να μας δώσουν να επιβάλλουν αντίπεινα μέτρα αντίπεινα αυτές οι χώρες γιατί ό,τι κακό μπορούσαν να κάνουν το έχουν ήδη κάνει σε αυτό το τομέα. Ευχαριστώ. Um, Η κυρία Βάλερ θέλει να δευτερολογήσει, όμως θέλω να ακούσω και την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Ε, να ακούσουμε πρώτα λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά να δώσω το λόγο και στην κυρία Βάλερ και στον κύριο Έγγελ. Δεν ξέρω ποιον, ποιος θέλει να λάβει το λόγο, κύριε Πίρενς, κύριε Γέρσεν, κάποιος από τους δυο σας. Θα ήθελα να ακούσω πρώτα από την πλευρά του εμπορίου και μετά να δούμε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Μπαλτασάρε που μας θυμήσατε το ιστορικό αυτής ε, της ε, αυτή, αυτού του, ε, αυτής της πρότασης. Έχουμε προβλήματα πρόσβασης ε, στις ε, ξένες αγορές και δεν πρέπει να χάνουμε την προοπτική στη συζήτησή μας. Αυτό που προτείνω να κάνουμε και συγγνώμη που άργησα κιόλας, αλλά από ό,τι κατάλαβα περισσότερο επικεντρώνεται η συζήτηση στην εκτίμηση επιπτώσεων που εκπώνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χθε είχαμε τη δυνατότητα να ε, πούμε ήδη κάποια πράγματα. Είναι ένα πολύ πυκνό και περιεκτικό κείμενο. Υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει να τα εξετάσουμε πολύ προσεκτικά, αλλά ένα ε, πράγμα που μας εξέπληξε ε, πρώτο ήταν ε, μια σοβαρή διαφορά μεθοδολογίας που είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να το αναφέρω σήμερα γιατί ίσως είναι η βασική συζήτηση που πρέπει να κάνουμε πριν μπούμε στην εκτίμηση των πολιτικών που προτείνει η πρόταση. Στην εκτίμηση επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προσπαθήσαμε και νομίζω ότι αυτό αναγνωρίστηκε και από τις μελέτες του Κοινοβουλίου ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο σε αυτό το τομέα να συλλέξει κανείς πολύ καλά δεδομένα γιατί πρώτον υπάρχουν ε, ακόμη και μεταξύ των ε, μερών ε, DPA υπάρχουν πολύ διαφορετικοί τρόποι συλλογής των δεδομένων και είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα όταν βγαίνει κανείς από τις χώρες που συμμετέχουν στις ε, συμφωνίες ε, προμηθειών. Ε, βασιστήκαμε στις δεσμεύσεις, στις νομικές δεσμεύσεις των εταίρων μας που μας εξασφάλισαν πρόσβαση για τις επιχειρήσεις μας υπό συγκεκριμένους όρους. Αυτό είναι αυτό θα ήθελα να πω. Δεν είναι μία προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μόνο μισό λεπτό να απομακρύνω το κινητό μου, είναι κάτι το οποίο ε, δεν το εφήβραμε μία νυχτή. Ε, είναι μία προσέγγιση την οποία ακολουθεί κατά κάποιο τρόπο και ο ΠΟΕ. Και αναφέρομαι σε μία έκθεση, την οποία επίσης παραθέσαμε χθε. Υπάρχει μία έκθεση του ΠΟΕ το από το 2011 για την αξιολόγηση της ε, μελλοντικής ε, προσχώρησης ε, κρατών στον ΠΟΕ σε σχέση με τις δημόσιες συμβάσεις. Αυτό, αυτό δείχνει ακριβώς τις ευκαιρίες ανοίγματος αγορών βάσει των συμφωνιών που έχουν συναυθεί και κάνει τη διάκριση μεταξύ από τη μία ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά και από την άλλη του βαθμού δίσδυσης στις αγορές. Η μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξετάζει αντιθέτως ε, το ποσοστό διείσδυσης στις αγορές και νομίζω ότι κάποια από τα συμπεράσματά σας, αν ακολουθήσει κανείς αυτόν τον, ε, αυτή την εναλλακτική λύση, ε, μπορεί να υπάρξουν κάποια κίνδυνοι. Στην ίδια μελέτη ΠΟΕ παράλληλα με μια μελέτη που έγινε από τη Γενική Διεύθυνση Μάρκτ πριν από μερικά χρόνια για την Ευρωπαϊκή Ένωση, επισημαίνει κάτι σημαντικό. Όταν βλέπει κανεί τα κέρδη πρόσβασης αγοράς, δεν πρέπει να ε, προσμέτρα κανεί μόνο αυτά σε σχέση με τις διασυνοριακές πωλήσει, όχι μόνο δηλαδή να βασίζεται στι διασυνοριακές πωλήσει, ε, ε, δηλαδή την πρόσβαση ξένων ε, εταιριών στην Ευρώπη, αλλά πρέπει να δει κανεί και τις θηγατρικές εταιρείε, δηλαδή κατά πόσο υπάρχει μια ε, παρουσία των εταιριών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δει κανεί την αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή έχουμε ένα πολύ ανοιχτό σύστημα επενδύσεων, οι περισσότερες ξένες εταιρείε που συμμετέχουν στις δημόσιες προμήθειες τις δικές μας, το κάνουν μέσω θηγατρικών με έδρα την Ευρωπαϊκή Ένωση, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει λοιπόν μεγάλο ποσοστό επιτυχίας, ε, κάτι το οποίο ήταν ε, συγκρίσιμο και δεν υπήρχε τελάξ, τεράστια διαφορά μεταξύ του αν ήταν κανείς ένας ε, εγχώριος ή ένας ξένος προμηθευτής. Αυτό ε, μας βάζει σε μια διαφορετική κατηγορία σε σχέση με, τους, ε, με, τα, υπόλοιπα ε, συμβαλόμενα μέρη. Γιατί οι υπόλοιποι έχουν πολύ περιορισμένες επιλογές, πολύ περιορισμένες δυνατότητες ξένων επενδύσεων. Αν δει κανεί τα πορίσματα της μελέτης της, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ένα από τα συμπεράσματα τα οποία μου έκανε πολύ εντύπωση είναι ότι ο παράγοντας ανοίγματο στη Ρωσία, ε, στην Ινδία ε, και στην Κίνα ε, είναι συγκρίσιμος με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν να ισχύει ε, γιατί οι ευρωπαϊκές εταιρείες, αν δει κανείς ε, τα στοιχεία του ΩΣΑ σε σχέση με το πόσο ανοιχτά ε, είναι αυτά τα κράτη για ξένες επενδύσεις, άμεσες επενδύσεις, είναι το ακριβές αντίθετο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που σημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείε πρέπει να προσπαθήσουν να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις χώρες μέσω διασυνοριακών συμβάσεων και επομένως ε, είναι σαν να συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Γιατί όταν βλέπει κανεί το ποσοστό διείσδυση, βλέπει μόνο το διασυνοριακό κομμάτι τη εξίσωση. Οι επιχειρήσει μα είναι υποχρεωμένε να λειτουργούν έτσι. Οι περισσότερες ξένες εταιρείες είναι πολύ ευκολότερο να εγκατασταθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όταν λειτουργούν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ταξινομούνται και χαρακτηρίζονται ω ευρωπαϊκέ εταιρείε. Και αν δεν μιλούμε για ποσοστά ε, δεν ε, το λαμβάνουμε αυτό υπόψη. Οπότε ένα μεγάλο κομμάτι κομμάτι του υπολογισμού δεν το λαμβάνετε υπόψη όταν βλέπετε πόσο δραστήριες είναι οι ε, ξένες εταιρείε στην ευρωπαϊκή αγορά. Και αυτό το λέω σε σχέση με τη μελέτη του ΠΟΕ ε, και ευχαρίστω να σας τη διαθέσουμε αν θέλετε. Κάτι ακόμη, μια πρόταση στην εκτίμηση επιπτώσεων ήταν ε, η απειλή ε, περισσότερων δυσκολιών ε, για την πρόσβαση στις ξένες αγορές και ότι αυτό είχε διωγγωθεί κάπως. Υπάρχει μια αυξανόμενη τάση για χώρες, κάποιες χώρες να έχουν πιο εθνική πολιτική σε σχέση με τις δημόσιες συμβάσεις ε, τα περισσότερα συμβαλόμενα μέρη όχι μόνο ακολουθούν τέτοια μέτρα, αλλά τα επιβάλλουν κιόλα. Κάτι το οποίο αναφέρεται στο έγγραφο του ΠΟΕ. Και το λέω αυτό για να σα πω και πάλι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν, βλέπει, δεν είναι η μόνη που βλέπει προβλήματα στον ορίζοντα και άλλοι διεθνεί οργανισμοί βλέπουν την ίδια τάση και εκφράζουν τι ίδιε ανησυχίε για το πού πηγαίνουμε. Ε, υπάρχουν λοιπόν κάποια μεθοδολογικά ζητήματα τι μετρά κανείς, το ποσοστό διείσδυση, όπω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η μελέτη του, μπορεί να είναι ένα ενδιαφέρον δείκτης για το πόση επιτυχία έχει κάποιο διασυνοριακά. Είναι ενδιαφέρον, αλλά είναι ενδιαφέρον μόνο αν ε, τη διασυνοριακή πρόσβαση προσμετρά κανεί. Δεν λαμβάνει υπόψη αυτά που πρέπει να συμπεριλάβουμε στην αξιολόγηση αν θέλουμε να έχουμε μια πλήρη εικόνα του πόσο δραστήριε είναι οι ξένε εταιρείε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τότε πρέπει και τι θηγατρικέ των ξένων εταιριών να τι λάβουμε υπόψη. Και είναι τεράστια διαφορά σε αυτή την περίπτωση για την ευρωπαϊκή αγορά, γιατί ε, είναι πολύ πιο εύκολο για μια ξένη χώρα να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν υπάρχει και διάκριση αυτή τη στιγμή υφίσταται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η βασική μεθοδολογική διαφορά και νομίζω ότι πραγματικά είναι παράξενα αυτά τα αποτελέσματα και θα ήταν δύσκολο κανείς όντως να αποδεχθεί ότι η Κίνα και η Ρωσία είναι ε, σε συγκρίσιμο βαθμό ανοιχτέ με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την προσφασιμότητα των ξένων εταιριών στι αγορέ του. Και πραγματικά, αν λάβουμε αυτό ω βασική υπόθεση, θα ήταν μάλλον περίεργο. Δεν ξέρω αν ο συνάδελφο από τη Γενική Διεύθυνση Μάρκ θέλει να πάρει το λόγο. Απλώ λίγο σύντομα, λέει ο πρόεδρο, γιατί έχουμε αργήσει. Θα ήθελα απλώ να πω ναι, να μας στείλετε όλα αυτά τα στοιχεία, τα λεπτομερή που έχετε. Είμαι σίγουρος ότι και ο εισηγητής μας τα θέλει πρέπει να περάσουμε στο επόμενο θέμα, οπότε πάρα πολύ σύντομα παρακαλώ. Mm. Ευχαριστώ πολύ. απλώς να επιβεβαιώσω ότι στο πλαίσιο αυτό είναι δύσκολο να συλλέξει κανείς δεδομένα στην εσωτερική αγορά. Είναι ακόμη πιο δύσκολο αν θέλει να έχει κανείς ε, ε, ε, σαφέστερα και ακριβέστερα στοιχεία σε ευρύτερο πλαίσιο ε, και μιλάω βέβαια για κάτι που αφορά και τρίτες χώρες. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν ε, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι δυνατόν ε, να έχουμε μία πλήρη αξιολόγηση ε, διαφορετικών πραγμάτων ε, υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Πρώτον, υπάρχει αυτό το θέμα της εκτίμησης επιπτώσεων από τους εμπειρογνώμονες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρόσφατα το λάβαμε, όπως είπαμε και στην Ίντα, θα το εξετάσουμε και πάλι. Και δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο να ε, λέμε ότι όλες, ε, όλα τα στοιχεία που αναφέρουν αυτά, αυτοί οι εμπειρογνώμονες είναι ακριβώς ίδια. Αν, δει, αν εξετάσει κανείς καλύτερα, ε, θα δει ότι υπάρχουν διαφορετικού είδους αξιολογήσεις που γίνονται στις διάφορες μελέτες. Όσον αφορά το σχέδιο γνωμοδότησης ε, του κυρίου Έγγελ, το γεγονός ότι αναφέρεται στην ανάγκη ύπαρξης ε, συνέπειας μεταξύ ε, των διαπραγματεύσεων στην αθεώρηση των οδηγιών και και κάποιες άλλες ρήτρε ή αντίστοιχες ρήτρε είναι βέβαια πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως θέλουμε να λάβουμε κάτι τέτοιο υπόψη. Μάλιστα. Δεν έχουμε χρόνο. Ε, Φρανκ Έγκελ, έχεις να προσθέσεις τίποτα? Κι εγώ δεν έχω χρόνο. Μάλλον δεν έχω και επαφή με τα πράγματα. Αναγνωρίζω βεβαίως αυτά τα οποία είπαν ε, οι συνάδελφοι, τα σημειώνω. Μπορεί να έχει νόημα να ε, πείσουμε, στείλουμε πίσω την πρόταση, γιατί δεν νομίζω να βγαίνει και τίποτα καλό. Δεν νομίζω ότι είναι μια πρόταση που δίνει πάρα πολλέ προοπτικέ. Να δούμε τέλο πάντων, ε, να περιμένουμε και τι τροπολογίε των ε, συναδέλφων. Να δούμε και θα δούμε κατά πόσο μπορούμε να το λάβουμε υπόψη ως πρόταση στην ε, καθήλυνα αρμόδια επιτροπή. Θα δούμε τι θα γίνει. Ευχαριστώ πολύ που εγκρίνετε ε, αυτό που προσπαθώ να κάνω. Καλώς. Προφανώς συνδεόμαστε τις εργασίες της ΣΥΝΤΑ και θα συζητηθεί και θα συνεχιστεί η συζήτηση και για την οδηγία για τις κρατικές προμήθειες την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, προθεσμία για τροπολογίες είναι 11 Ιουλίου και από εκεί πέρα βλέπουμε. Προχωράμε. Ελπίζω να έχουμε μέχρι τότε κάποιες, ε, κάποιες ειδήσεις όσον αφορά την οδηγία για τις ε, δημόσιες προμήθειες μέχρι τότε. Ευχαριστώ όλους, ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάμε στο επόμενο σημείο που είναι το τελευταίο. Ήταν ε, δύσκολη ψηφοφορία το πρωί. Καμιά φορά η εγκρίση όσον αφορά για τις πολύ σε ευρωπαϊκό επίπεδο η διαφορά ήταν πολύ μικρή στις ε, ψήφους. Ο Hans Peter και η κυρία Γκέπαρτ να μας πούν κάτι για τις τροπολογίες, να σχολιάσουν και σκιώδεις. Υπήρξαν επαφές με τους σκιώδεις. Περιμένουμε να διεξαχθεί μια περίπλοκη διαδικασία στο θέμα. Ε, καλωσορίζω τον κύριο Στέρ Μαέρ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τακτικός συνομιλητής μας. Ο κ. Κρόιτσμαν είναι εδώ από τους Κιώδης, ο κ. Ρούλε, ο κ. Φόξ ελπίζει να καταφτάσει. Είναι στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, όπου συζητείται έκθεσή του. Ποιος θα ξεκινήσει. Κυρία Γκέπχαρτ, ο κ. Μάιερ. Κυρία Γκέπχαρτ σήμερα το πρωί. Είχαμε συμφωνήσει εναλλακτικά να το κάνουμε ο Χανς Πέτερ είχε ξεκινήσει, ας ξεκινήσω εγώ σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, εντάξει, σήμερα θα συζητήσουμε για τις τροπολογίες. Καθίσαμε με τους σκιώδεις εισηγητές και τα είδαμε και στις σκιώδεις εισηγήτριες. Κάποιοι ήταν παρόντες και παρούσες, όχι όλοι. Διαπιστώσαμε ότι μεταξύ των δύο θέσεων αρχής που έχουμε μπροστά μας δεν είναι εύκολο να υπάρξουν συμβιβαστικές λύσεις, συμβαστικές προτάσεις. Ή θα ακολουθήσουμε την πρόταση Μάιερ ή την πρόταση Γκέπαρτ. Μεταξύ των δύο προτάσεων δεν είναι εύκολο, δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν συμβιβασμοί. Επειδή είναι τελείως διαφορετικές προτάσεις η μία από την άλλη. Γι' αυτό δεν έχουμε συμβαστικές τροπολογίες μπροστά μας. Γιατί δεν είναι εφικτό να επιτευχθούν τέτοιες συμβαστικές τροπολογίες. Στη συνεδρίαση μετά στη συνέχεια συζητήσαμε για το πώς θα συνεχίσουμε, ποια διαδικασία θα ακολουθήσουμε. Και φυσικά ο Hans Peter από πλευράς του κάποιες τροπολογίες συμβιβαστικές με άλλους θέλει να προετοιμάσει, όπως και εγώ θέλω να προετοιμάσω κάποιες συμβαστικές τροπολογίες με άλλους συναδέλφους. Δεν έχουν ολοκληρωθεί όμως αυτές ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη. Και έτσι δεν τις έχουμε ούτε αυτές στα χέρια μας σήμερα. Έχουμε όμως μία απόφαση επί θέματος αρχής που λάβαμε, ότι φυσικά ανάλογα με το ποια κατεύθυνση θα θελήσουμε να ακολουθήσουμε στην αρχή της ψηφοφορίας, φυσικά πρώτα η τροπολογία Νίμπλερ Weisgerber θα τεθεί σε ψηφοφορία, σε ψήφιση, που λέει δεν θέλουμε κανονισμό ούτε οδηγία, επαναπομπή απλά ίσια και κατευθείαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λέμε όμως ότι όπως έχουν οι πλειοψηφικές ε, ε, αναλογίες δεν θα υπάρξει πλειοψηφία. Μια και ούτε το ΕΛΚ, ούτε οι φιλελεύθεροι, αλλά και ούτε και οι σοσιαλδημοκράτες, δεν ξέρω τι γίνεται με άλλες ομάδες, στον πίνακα ψηφοφορίας δεν θα βάλουν ένα θετικό πρόσημο, δεν θα βάλουν ένα συν για να υπερψηφιστεί κάτι τέτοιο, καθότι γνωρίζω τουλάχιστον. Στη συνέχεια θα ληφθεί απόφαση για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουμε. Σημαντικό θέμα η γραμμή Μάιερ ή η γραμμή θα εγκριθεί και θα ακολουθηθεί. Και ανάλογα με το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, μια ολόκληρη σειρά τροπολογιών θα έχουμε που θα καταπέσουν ή από τη μία κατηγορία, από τη μία όχθη, από τη μία πλευρά ή από την άλλη, ανάλογα με το ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσουμε. Και έτσι θα έχουμε τις επισημάνσεις στον κατάλογο, στον πίνακα ψηφοφορία σχετικά. Μετά έχουμε και μια σειρά τροπολογιών που αφορούν το ένα σύστημα που όμως και μπορούν να γίνουν δεκτές και από το άλλο σύστημα, από την άλλη πλευρά. Σκεφτήκαμε αν θα έχουμε ένα σύστημα συμβαστικών τροπολογιών που θα μπορούσαμε να εκπονήσουμε. Διαπιστώσαμε όμως ότι είναι υπερβολικά περίπλοκο κάτι τέτοιο και γι' αυτό υπό τη μορφή προφορικών τροποποιήσεων θα ε, καταθέσουμε προτάσεις εκεί όπου είναι αναγκαίο να γίνει κάτι που θα αναφέρονται στον πίνακα ψηφοφορίας ώστε με πλήρη διαφάνεια να μπορέσουν όλα αυτά να διευθετηθούν ψηφίζοντας. Και έτσι συμφωνήσαμε μεταξύ των κοινοβουλευτικών ομάδων, τουλάχιστον μεταξύ αυτών που ήταν παρούσες ως ομάδες, να μην έχουμε ε, διαφωνία σε αυτές τις προφορικές τροποποιήσεις που θα κατατεθούν να μην έχουμε ενστάσεις και αντιρρήσεις. Θα ρωτήσουμε όμως και εκείνες τις κοινοβουλευτικές ομάδες που δεν ήταν παρούσες αν συμφωνούν με αυτή τη διαδικασία. Μια και δεν έχουμε συμβαστικές τροπολογίες που θα προετοιμαστούν ώστε αμοιβαία λοιπόν να μπορέσουμε να έχουμε συμφωνήσει κάτι, να μην υπάρξουν ελιγμοί και χειραγωγίες, ε, χειραγωγήσεις επ' αυτών, διότι είναι πολύ περίπλοκα θέματα και να, δεν θέλουμε να είμαστε αντιπαραγωγικοί, θέλουμε με διαφάνεια να εργαστούμε. Αυτά είναι αυτά τα οποία θέλω να σας αναφέρω τώρα. Επακούμε σε αυτά. Αν υπάρχει κάποια επιθυμία κάτι να συζητηθεί επί της ουσίας, μια και σήμερα δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό πιστεύω, μια και ο χρόνος πιέζει, εκτός αν ξεκινήσει ο Χάνς Πέτερ ή κάποιος άλλος με αυτά, τότε θα ξαναζητήσω τον λόγο ώστε επί της ουσίας να πω δύο λόγια για κάποια πράγματα. Επαρκούμε σε αυτά, ευχαριστώ. Καλώς κατανοώ ακριβώς τη θέση σας όσον αφορά συμβαστικές τροπολογίες. Πρέπει να κάνουμε κάποια ποιοτική δουλειά όσον αφορά τον κατάλογο ψηφοφορία και να δούμε ποιες είναι οι συγκεκριμένες θέσεις Επιτροπής και ποιες τροπολογίες συμπεριληφθούν, ποιες δεν θα συμπεριληφθούν, ποιες θα είναι οριζόντιες τροπολογίες, θα εμπίπτουν στις δύο προτάσεις. Σίγουρα μπορούμε να το καταφέρουμε. Ο κ. Μάιερ έχει το λόγο. ναι, ευχαριστώ πολύ αληθεύουν στην ουσία ουσιαστικά αυτά που μόλις είπε η Εβελίν Γκέπχαρτ επειδή στην αρχή χρειαζόμαστε μια απόφαση για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουμε. Αλλιώς δεν θα ξέρουμε τι θα ψηφίζουμε και προς πού θα πορευτούμε. Λοιπόν, πράγματι συζητήσαμε για τη δυνατότητα να έχουμε προφορικές τροποποίησεις που θα κατατεθούν η γραμματεία και ένα ηλεκτρονικό μήνυμα απέστειλε. Καλύτερο όμως είναι γραπτά να διατυπωθούν αυτά και όλα αυτά θα πρέπει γραπτά να είναι διαθέσιμα. Θα, έχει, θα έχουμε ένα σύμφυρμα, ένα συνονθήλευμα μεταξύ της ελευθερίας, ε, ελεύθερης δυνατότητας κατάθεσης τροποποιήσεων προφορικών με τις γραπτές προτάσεις που θα έχουμε. Μέχρι τώρα επτά συμβαστικές προτάσεις έχω εκπονήσει, που τις έχω στα γερμανικά όμως αυτές. Το δυνατόν πολλοί συνάδελφοι καλούνται να συμμετάσχουν που ανεξάρτητα από το θέμα απόφασης αρχής θα έπρεπε να συνεχίσουμε προς αυτή την πορεία διότι συνεχίζουμε την εξέταση σε πολλά επιμέρους θέματα και είναι λοιπόν σκόπιμο διασυνοριακά να εξεύρουμε συμβαστικές προτάσεις που θα, στις οποίες θα καταλήξουμε. Έξι προτάσεις από αυτές τροπολογίες είναι προσαρμογή του κειμένου ε, μία ε, συμβιβαστική πρόταση είναι με την συνάδελφο Ρέπο για την διατήρηση της ε, εθελούσιας δυνατότητας αυτού του μέσου και το, του πεδίου εφαρμογής. Όλα τα άλλα είναι τροποποιήσεις και συμβαστικές τροπολογίες. Και πέρα από αυτά έχω και τουλάχιστον για το δικό μου τομέα τέσσερις συναφείς περιορισμούς και όσον αφορά και κάποιους ορισμούς που θέλουμε να υιοθετηθούν. Παράδειγμα, ορισμός τι είναι η ε, σύμβαση ε, σε σχέση με τους καταναλωτές. Είναι κάτι διαφορετικό από κανονικές συμβάσεις ε, συναλλαγών. Πρέπει να καθορίσουμε όπως με το online fair δηλαδή τη διαδικτυακή σύμβαση συναλλαγής, να δούμε τι θα γίνει ατομικά μια και μια προσωπική επικοινωνία με email, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν είναι μια τέτοιου είδους σύμβαση καθαρά. Λοιπόν, πρέπει να υπάρξουν κάποιες αποσαφηνίσεις και κάποιοι προσδιορισμοί. Αυτή τη στιγμή τι μπορούμε να διαπιστώσουμε. Έχουμε δύο κατηγορίες προτάσεων και δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι υπάρχει αυτή η διαφορά, αυτός ο κατακαιρματισμός. Συνεχίζω να πιστεύω ότι πρέπει να είναι εθελούσιου χαρακτήρα αυτά τα μέσα. Είναι το καλύτερο που χρειαζόμαστε για να ανοίξουμε την αγορά. Διότι είμαστε Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτών. Πρέπει να διευρύνουμε την εσωτερική αγορά και δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό συμπληρώνοντας διαρκώς ε, νομοθετήματα μονομερός υπέρ των καταναλωτών. Αυτό δεν ανοίγει την εσωτερική αγορά ακολουθεί μια άλλη πορεία. Εμείς θέλουμε όμως να ανοίξουμε το πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς, να έχουμε την ευκαιρία πρόσβαση σε αυτήν παντού, με την καλύτερη προσφορά και το καλύτερο προϊόν που μπορούμε να αγοράσουμε σε αυτές τις συναλλαγές και για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να σκεφτούμε πώς θα μπορέσουμε να ανοίξουμε περισσότερο την εσωτερική αγορά, πόσο μπορούμε στη συνέχεια να προστατεύουμε τους καταναλωτές. Και στο τέλος τέλος τίποτα δεν είναι πιο λογικό και συνετό και συνεκτικό από το να υπάρξουν κάποιες ρυθμίσεις και διατάξεις ώστε να υπάρξει ένα υψηλότερο επίπεδο προστασίας καταναλωτών αλλά να μην έχουμε έτσι, ας το πω έτσι, περιοριστικό πλαίσιο των 28 κρατών μελών όσον αφορά την εσωτερική αγορά. Πρέπει να μεριμνήσουμε να είναι λογικά, λογικές οι αναλογίες των πραγμάτων και για την εσωτερική αγορά. Τα λέω αυτά διότι το Κοινοβούλιο αμφισβητείται ότι έχει τοποθετηθεί με κάθετο τρόπο για ένα εθελοντικού χαρακτήρα τέτοιο μέσο στην απόφαση του 2011, δύο χρόνια πριν δηλαδή. Και υπό το εδάφιο 5, τι αναφερόταν τότε, ότι το Ευρωκοινοβούλιο προτιμά την εναλλακτική λύση δυνατότητας 4, 4 <clears throat> με ένα εθελοντικού χαρακτήρα μέσο μέσω κανονισμού, μετά αποσαφήνιση της νομικής βάσης. Έχει αποσαφινιστεί η νομική βάση από την νομική υπηρεσία. Πιστεύει το Ευρωκοινοβούλιο ότι αυτό το εθελοντικού χαρακτήρα μέσα, μέσω, μέσω ενός toolbox, μέσω μιας εργαλειοθήκης, μέσω της διοργανικής συμφωνίας θα μπορούσε να συμπληρωθεί. Όχι να υποκατασταθεί, να συμπληρωθεί. Και υπό το σημείο 6 θεωρεί το Ευρωκοινοβούλιο ότι μόνο η μορφή ενός κανονισμού καθορίζει και δίνει τα αναγκαία πλαίσια και την αναγκαία νομική ασφάλεια. Και στο εδάφιο 7 επαναλαμβάνει και τονίζει το Ευρωκοινοβούλιο ότι η δημιουργία μέσω νομικού πλαισίου μιας τέτοιας ε, ε, δυνατότητας δίνει προτερήματα στις επιχειρήσεις, μείωση των δαπανών και του κόστους και στους καταναλωτές προσφέρει νομική βεβαιότητα και ασφάλεια, προστασία καταναλωτών και τα νομικά συστήματα στα επιμέρους κράτη-μέλη που δεν θα ασχολούνται με θέματα αλλοδαπού δικαίου, αλλά θα επαρκούνται στη λειτουργία τους ώστε να έχουμε μια καλύτερα λειτουργούσα ενιαία εσωτερική αγορά. Αυτή είναι η μεγάλη απόφαση. 421 υπέρ, 145 εναντίον και 8 αποχές. Αυτή ήταν η απόφαση τότε που είχαμε λάβει. Δεν μπορούμε να αμελήσουμε, να αγνοήσουμε αυτή την απόφαση και γι' αυτό πιστεύω ότι είμαστε στη σωστή πορεία αν με το εθελοντικού χαρακτήρα μέσω συνεχίσουμε την πορεία μας. Θέλω να περιοριστεί το πλαίσιο αυτό και σε σχέση με τις συμβάσεις στο ηλεκτρονικό ε, εμπόριο αυτό είναι το κυριότερο θέμα που πρέπει να ρυθμίσουμε Εξειδικευμένα λοιπόν για αυτό το μέσο των ε, ηλεκτρονικών συμβάσεων πρέπει να προβλέψουμε και να μεριμνήσουμε για το άνοιγμα της εσωτερικής αγοράς και για την προστασία των καταναλωτών. Έτσι θα έχουμε καταφέρει κάτι το εποφελές. Ευχαριστώ. Κύριε Κυρία Γκέπχαρτ, θέλει να παρέμβει εκ νέου. Θα κάνουμε ένα γύρο παρεμβάσεων των σκιωδών και μετά να ακούσουν κάποιου Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ολοκληρώνουμε στο τέλο. Κύριο Κρόιτσμαν, καλωσορίζω και τον κύριο Φόξ. Δεν χρειάζεται να διαβάσω λοιπόν τις σημειώσεις του. Η κυρία Ρούλε δεν είναι εδώ και ο Σκρότσμαν πρώτος. Λοιπόν, εμείς εξακολουθούμε να λέμε ότι είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πείραμα αυτό με την προσφορά αυτή που γίνεται. Θα έπρεπε να μην υπερβάλλουμε και να μην υπερβαρύνουμε υπερβολικά αυτό το, αυτή την πρωτοβουλία για να μπορέσει να είναι λειτουργική. Θέλουμε, δεν θέλουμε να καταργήσουμε δικαιώματα καταναλωτών. Όταν θέλουμε, ξέρουμε ότι έχει μια φιλόδοξη πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τότε θα πρέπει και τα δικαιώματα των καταναλωτών να λαμβάνονται υπόψη. Δεν θα πρέπει να υπερβάλλουμε υπερβολικά όμως, ε, να μπορέσουν να ε, λειτουργήσουν όλα αυτά, γιατί διαφορετικά δεν θα έχουμε θετικό αποτέλεσμα και θα έχουμε περιορισμένη εμβέλεια βλέπουμε ότι η μεγαλύτερη πρόσθετη αξία θα ήταν η εσωτερική αγορά που μπορούμε να την αναπτύξουμε περαιτέρω και να την ανοίξουμε περισσότερο. Γι' αυτό για όσα, είπε, για όσα αναφέρονται από πλευρά του συναδέλφου Μάη θα δούμε τι θα κάνουμε τελικά με την ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Mr. Fox. Fox. Thank you, President. Sorry, just clearing... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ξέρουν οι συνάδελφοι ότι προτιμώ την προσέγγιση της κυρίας Γκέπαρτ στο θέμα αυτό διότι παρούσα πρόταση το δυνητική ευχέρεια εργαλείο θα είναι επιβαρυντικό και για την προστασία των καταναλωτών και για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Είμαι ανοιχτή στι δικέ σα προτάσει. Πρέπει να εξασφαλίσουμε την εφαρμογή των συμπεφωνημένων νομοθετημάτων, όπω την οδηγία του δικαιώματο των καταναλωτών χρησιμοποιώντας την οδηγία για τα νομικά εκέγγυα που υπάρχει ήδη και να εφαρμόσουμε και την οδηγία την ελάχιστη εναρμόνιση. Να πω κάτι που αφορά ειδικά το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι τροπολογίε που υπέβαλα που αφορούν τα άρθρα 106 και θα ζητούσα την κυρία Κέπχαρτ να τα λάβει υπόψη αυτά. Η δική τη προσέγγιση του κ. Μάγερ θα άφηνε του κατανοητέ του Ηνωμένου Βασιλείου με χαμηλότερο επίπεδο προστασία από αυτό που απολαμβάνουν τώρα. Με την τη νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, του Ηνωμένου Βασιλείου με την νομοθεσία, οι καταναλωτέ μπορούν να τερματίσουν τη σύμβαση εντό συγκεκριμένης περίοδου από την παράδοση αν δεν πληρούν τις συμβασιακές υποχρεώσεις. Είναι η βραχυπρόθεσμο, η δικαίωμα απόρριψη αποκαλείται. Και υπάρχει και ένα σύστημα σε διάφορα επίπεδα. Μπορεί να ζητήσει αντικατάσταση του προϊόντος ή επισκευή του προϊόντος και μετά να τεθεί τέρμα στη σύμβαση ή να ζητήσει επιστροφή χρημάτων αν τα αγαθά εξακολουθούν να μην α, ε, λειτουργούν σωστά και να μην πληρούν τις ε, προδιαγραφές. Τα δύο συστήματα είναι εναλλακτικά και δίνουν στον καταναλωτή επιλογή, δυνατότητα επιλογής. Μα διαλέξει σύστημα που θα ακολουθήσει. Ξεκαθάρισα βέβαια ότι προτιμώ την προσέγγιση Ιας Γκέπχαρτ, αλλά και η δική της και του κ. Μάιερ, αν επιλεγεί Κάποια από τις δύο, σε οποιαδήποτε περίπτωση εγώ θέλω να εξασφαλίσω τη σωστή προστασία των καταναλωτών του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν θέλω να μειωθεί το επίπεδο προστασίας των καταναλωτών του Ηνωμένου Βασιλείου. Καλός. Άλλος που επιθυμεί να παρέμβει. Ο κ. Στανεμάιερ. Τι άποψη έχει. Θέλετε να μιλήσετε πρώτη πριν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρία Γκέπχαρτ. Σας δίνω το λόγο τώρα. Ε, Σας ευχαριστώ. Στην αρχή περιορίστηκα μόνο να αναφέρω αυτά που είχαμε συμφωνήσει. Αλλά μια και οι συνάδελφοί μου τοποθετήθηκαν επί της ουσίας, πιστεύω ότι και εγώ επί της ουσίας θα έπρεπε να ξανατοποθετηθώ, ώστε όσοι μας παρακολουθούν να ξέρουν τι γίνεται μέσω του διαδικτύου. Να μάθουν περί τίνος πρόκειται. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Καταρχήν λοιπόν πρώτα, θα ήθελα με κάθετο και σαφή τρόπο να πω ότι εγώ με κανέναν τρόπο δεν θέλω την εσωτερική αγορά εις βάρος των καταναλωτών και των δικαιωμάτων τους να την ανοίξουμε. Το πρώτο μας και κυριότερο έργο είναι να μεριμνήσουμε το υψηλότατο επίπεδο προστασίας καταναλωτών που έχουμε στα κράτη-μέλη αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να μην αποδυναμωθεί, να μην υπονομευθεί. Και γι' αυτό θέλω να πω στον συνάδελφο ότι με κάθε σαφήνεια, δεν ξέρω το νομικό πλαίσιο πώς έχει σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν κάτι υποβληθεί που θα σημαίνει πρόσθετη αξία για το Ηνωμένο Βασίλειο, θα πρέπει να ε, δούμε ότι δεν είναι δυνατόν να υπονομεύεται μέσω ευρωπαϊκού, δικτύου, ε, ευρωπαϊκού δικαίου το εθνικό δίκαιο και λέτε εσείς ότι θα είναι λέει κάτι ενδιαφέρον αυτό πείραμα κύριε Κρότσμαν αλλά στην προστασία καταναλωτών δεν πρέπει να κάνουμε πειράματα πρέπει να μεριμνήσουμε παρέμβαση χωρίς μικρόφωνο πρέπει να μεριμνήσουμε και να διασφαλίσουμε ότι ένα υψηλότατο όσο δυνατόν υψηλότερο επίπεδο προστασίας καταναλωτών θα διασφαλίζεται και το ξέρετε ακριβώς κύριε Κρότσμαν λέτε κάτι πράγματα χωρίς μικρόφωνο ως παρατηρήσεις ε, Ξέρετε ότι στις διαπραγματεύσεις με τους επιχειρηματίες έχουμε σε σχέση με τους καταναλωτές την πιο αδύναμη θέση. Όταν προτείνεται κάποιο εθελοντικού χαρακτήρα σχήμα, μετά τι γίνεται, δεν έχουν άλλες ευκαιρίες οι καταναλωτές από το να δεχτούν αυτό που τους προσφέρεται όταν έχουν κάποια σύμβαση ή αγοράζουν κάποιοι, κάποιοι κάτω κάτι. Με αυτή την πρόταση λοιπόν θα είχαμε αποδυναμωμένη προστασία καταναλωτών. Δεν θέλουμε να γίνει κάτι τέτοιο. Και ένα χρόνο πριν από τις ευρωεκλογές να στείλουμε ένα τέτοιο πολιτικό μήνυμα στους πολίτες μας γυναίκες και άνδρες ότι θα αποδυναμωθεί το επίπεδο ε, προστασίας τους ως καταναλωτών δεν θέλουμε να γίνει κάτι τέτοιο και για ένα πράγμα θα ήθελα να πω τούτο για αυτό το οποίο έγινε και ψηφίσαμε το 2011 στην Ολομέλεια στο Ευρωκοινοβούλιο για αυτό το θέμα το 2011 πρέπει να πω ότι είναι κάτι που σε σχέση με την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων γύρω την κατηγορία, την επίκριση ότι σε τέτοιες σημαντικές αποφάσεις που λαμβάνονται από την Ολομέλεια ακολουθήθηκε μια πορεία χωρίς να ενημερωθούν όλοι οι ευρωβουλευτές για το πόσο φλέγον ήταν το θέμα και η εμβέλειά του. Διότι αν είχε γίνει κάτι τέτοιο θα είχαμε μια εντονότατη συζήτηση για αυτά τα θέματα τότε. Και τουλάχιστον όταν έχουμε αυτό το ψήφισμα το οποίο αναφέρεται τότε το σύνολο της πρότασης ψηφίσματος θα πρέπει να αναφέρεται και να φωτίζεται και να μην αγνοούμε ότι υπάρχει ένα σημείο 36, ένα εδάφιο 36 σε αυτό το ψήφισμα όπου λέγεται και σας το διαβάζω ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη να ελέγξει την ποιότητα και τα προϊόντα αυτά με τέτοιο τρόπο αν, για να διαπιστωθεί αν τα μέσα τα οποία προτείνονται μέσω του συμβατικού δικαίου για τέτοιου είδους συμβάσεις αγοράς λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες και τα συμφέροντα των καταναλωτών επιπρόσθετα για την προστασία τους για, και πέρα από την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς να διευκολύνονται οι συναλλαγές. Και η μελέτη επιπτώσεων που έχουμε και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η αξιολόγηση από τις επιμέρους υπηρεσίες που έχουμε στη διάθεσή μας δείχνει ότι ακριβώς αυτά τα σημεία δεν είναι διασφαλισμένα και δεδομένα δεν υπάρχει κάτι το πιστικό όσον αφορά αυτές τις συναλλαγές και το κόστος συναλλαγών όσον αφορά τις επιχειρήσεις. Γιατί επ' αυτών δεν υπάρχουν θέματα. Και όταν λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι χρησιμοποιήσαμε τα στοιχεία που είχαμε στη διάθεσή μας, ναι αλλά αν αυτά τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν δεν τοποθετούνται επ' αυτών των προβλημάτων, δεν μπορεί να υπάρξει μελέτη επιπτώσεων για τη συνέχεια διαπιστώσαμε ότι το όφελος για τους καταναλωτές είναι ελάχιστο, ελαχίστου επίπεδου, διότι αυτά που υποσχέθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκονται μεταξύ 0,4-0,7%. Σε αυτό κυμαίνονται. Αυτό δεν είναι προτέρημα και προστασία για τους καταναλωτές και νομίζω ότι και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Και γι' αυτό πολύ καλά και ωραίο ότι ελήφθη μία απόφαση το 2011 τότε, αλλά όμως ε, δεν βρίσκεται σε σταθερά θεμέλια, είναι σε σαθρά θεμέλια. Και αυτό το επιβεβαιώνουν οι υπηρεσίες μας. Και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο δεν ήταν δυνατόν για αυτή την μελέτη επιπτώσεων των επιπτώσεων ακόμα και από τους υπέρμαχους του συστήματος εθελοντικού χαρακτήρα δεν αναφέρεται, έχει αποσιοποιηθεί. Και αυτό είναι ο λόγος ότι, για τον λόγο του ότι η μελέτη επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι, δεν είναι σταθερή και αξιόπιστη. Ευχαριστώ. Παρακολουθώ μεγάλο ενδιαφέρον τη συζήτηση. Δεν θέλω να επαναληφθεί όμως η συζήτηση. θα έχουμε και άλλη δυνατότητα να διεξάγουμε τη συζήτηση μαζί με τον κύριο Κρόιτσμαν και η ομάδα του κύριο Κρόιτσμαν θα πρέπει να αποφασίσει κατά πόσο θα υποστηρίξουν την επιλογή. Εμείς θα έχουμε συζήτηση για ποια γραμμή θα ακολουθήσουμε. Θα τα αφήσουμε μέχρι την ψηφοφορία που θα προηγηθεί ψηφοφορία ψηφοφορία και από συζήτηση. Ήθελα να δώσω μερικά λεπτά στο κύριο Στέκεμα. Είναι 12.25 και λυπάμαι ότι έχουμε στριμωχθεί λόγω της ψηφοφορίας χρονικά. Ε, είδατε λοιπόν τις τροπολογίες. Έχετε συγκεκριμένα σημεία που αφορούν τις τροπολογίες. Δεν θέλω να δικαιολογήσετε τη θέση σας, την ακούσαμε επανειλημμένα, κάτω παρελθόν. Αλλά για τις τροπολογίες που θα επηρεάσουν ε, τη θέση σας. Αυτές ίσως να σχολιάσετε πριν κλείσουμε μέχρι το απόγευμα και μετά πρέπει να ετοιμαστούμε και για την ψηφοφορία της επόμενης εβδομάδας. Εκτός λοιπόν. μικροφών. Σχόλιο. Ο κύριος Μάιερ θα έχει δυνατότητα να μιλήσει ξανά. Εφόσον έκανε τον κόπο να έρθει κύριος ο Μάιερ, ας του δώσουμε τη δυνατότητα να σχολιάσει τις τροπολογίες, που είναι και το σημαντικότερο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η μεγάλη αντίθεση μεταξύ αυτών των δύο προσεγγίσεων είναι το θέμα του εθελοντικού χαρακτήρα μέσου ή μιας οδηγίας. Και με αυτή την ευκαιρία δεν θέλω να μακρηγορήσω. Ακριβώς η εθελοντική πλευρά δημιουργεί μια win-win situation, μια κατάσταση αμοιβαίου ωφέλους με μικρές δαπάνες να μπορούν αυτά τα προϊόντα να διοχετεύονται στην εσωτερική αγορά και οι καταναλωτές να έχουν μεγαλύτερη επιλογή από τέτοιου είδους ευρύτερη προσφορά προϊόντων και αυτό είναι το όφελος για τους καταναλωτές και έχουμε προστασία καταναλωτών που θα είναι ίδια ή ανώτερη σε σχέση με το εναρμονισμένο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είναι ή ίσο το επίπεδο ή και ανώτερο με εκείνο το οποίο στα περισσότερα κράτη-μέλη ισχύει για τέτοια μέτρα τα οποία δεν έχουν εναρμονιστεί ή τουλάχιστον ξεπερνούν και την οδηγία εναρμονισμού. Δίνουμε λοιπόν και σε καταναλωτές και σε επιχειρήσεις μια επιλογή που δεν είχαν μέχρι σήμερα και δεν έχουν μέχρι σήμερα και αυτό είναι το θετικό για την εσωτερική αγορά και με μεγάλο ενδιαφέρον προσβλέπει να δει την ψηφίση αυτού του θέματος στην Επιτροπή σας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύντομα αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Κύριε Κρόιτσμαν, πολύ σύντομα. Δεν έχουμε χρόνο. Πάρα πολύ σύντομο σχόλιο. Ήθελα να πω στη συνάδελφο Γκέπαρτ, ας αφήσει την πάλη των τάξεων και τις αναλήθειες. Οι Γερμανοί πολιτές αγοράζουν ε, τα προϊόντα τους σύμφωνα με γερμανικό δίκαιο και με υψηλότατο επίπεδο προστασίας καταναλωτών. Και οι Βρετανοί και τα λοιπά το ίδιο και δεν αλλάζει τίποτα. Τι έχουμε εδώ, οι Λουξεμβούργοι, οι Λετονοί ή οι άλλοι αγοράζουν διασυνοριακά και το είπε αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν κάνουν κάτι τέτοιο θα έχουν ευκαιρία εταιρείες να επιλέγουν και να αγοράζουν προϊόντα από μια μεγάλη εσωτερική αγορά. Κανείς δεν υποχρεώνεται κυρία Γκέπαρτ, καμιά επιχείρηση να προσφέρει τα προϊόντα της. Και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε αυτή την κατάσταση και είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυξήσαμε το επίπεδο προστασίας καταναλωτών για να δοθούν κίνητρα για τους πελάτες που θέλουν να έχουν μια τέτοια ευκαιρία. Αυτό είναι όλο και όλο. Και όταν λέτε τώρα ότι θέλουμε να στραγγαλίσουμε την ε, προστασία καταναλωτών, ε, ε, δεν έχει κανένα νόημα με κάτι τέτοιο. Είναι αναλήθειες αυτά. Δεν ισχύουν, δεν ευσταθούν. Και το είχα πει ότι έχει μόνο τότε νόημα αυτά τα 28 συστήματα να μπορέσουν να λειτουργήσουν με τέτοιο τρόπο σωστά όταν οι επιχειρήσεις έχουν κίνητρα για να προχωρήσουν προς μια τέτοια κατεύθυνση. Αυτό είναι όλο και όλο να προσφέρουν τα προϊόντα τους στους αγοραστές, στους πελάτες. Οι καταναλωτές δεν είναι υποχρεωμένοι να αγοράζουν αυτά τα προϊόντα, μπορούν σύμφωνα με γερμανικό δίκαιο και σύμφωνα με γερμανικό δίκαιο προστασίας καταναλωτών να αγοράζουν ή οι Βρετανοί το ίδιο. Δεν είναι υποχρεωτικό να αλλάξει κάτι. Επαναλαμβανόμαστε νομίζω. Θα ήταν χρήσιμο να, είμαστε, να είχαμε ακούσει όλα αυτά τα ενθουσιώδη επιχειρήματα όταν είχαμε κάνει την ακρόασή μα πριν από μερικού μήνε. Τότε είχαμε πολύ αδύναμα επιχειρήματα, αλλά ίσω εξελιχθήκαμε με τον καιρό. Κοιτάξτε, εγώ το λέω επειδή κάθομαι εδώ ως ανεξάρτητος παρατηρητής και βλέπω συνεχώς ε, πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Να σας δώσω εσάς ε, το λόγο για να ολοκληρώσουμε τη συνεδρίαση, κύριε Μάγερ. Ναι, ευχαριστώ. Κάθε ένα μπορεί να τοποθετηθεί δύο φορές και αυτή είναι η δεύτερη τοποθέτησή μου. Δύο σημεία μόνο, Εβελίν Γκέπαρτ. Είπες, η ενιαία εσωτερική αγορά δεν πρέπει να ανοίξει εις βάρος των καταναλωτών. Δεν το βρίσκω σωστό αυτό, γιατί δεν αληθεύει, δεν είναι εις βάρος των καταναλωτών. Ανοίγει η εσωτερική αγορά σε τέτοιο βαθμό με τι πρόσθετε προσφορέ που θα γίνονται προϊόντων. Και μετά πρέπει να δεχτούμε όταν ως καταναλωτές αγοράζουμε κάτι δεδομένες ε, συνθήκες και δεδομένους όρους. Αλλά αυτό σε σχέση με τις δυνατότητες που ανοίγονται για αυτούς. Αυτή είναι η διαφορά μας μεταξύ μας. Εγώ θέλω οι καταναλωτές οι οποίοι δεν θα πηγαίνουν με εθνικό δίκαιο να αγοράζουν θα έχουν μια προσφορά προϊόντων πιθανότατα υπό ευρωπαϊκό δίκαιο, αλλά μπορούν να αγοράσουν αυτά τα προϊόντα. Τώρα δεν μπορούν να τα αγοράσουν προτού γίνει αυτό. Πρέπει να διευρύνουμε λοιπόν την αγορά, όχι εις βάρος των δικαιωμάτων καταναλωτών, αλλά καθιστούμε δυνατόν να υπάρξει μια προσφορά για να κινηθούμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Να μην δημιουργηθεί εντύπωση ότι όταν έχουμε εθελοντικό πλαίσιο εφαρμογής τέτοιων συμβάσεων δεν θα υπάρχει προστασία καταναλωτών. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, δεν ευσταθεί διότι αυτό το νομοθέτημα περισσότερο από το ίμιση των άλλων στις, ε, στις άλλες χώρες δίνει σε περισσότερο από 50% από αυτές υψηλότερο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. Ας μην είμαστε λοιπόν, ας το πω έτσι, ισοπεδωτικοί στις τοποθετήσεις μας. Ευχαριστώ. Προφανώ θα το συζητήσουμε πολλέ φορέ ακόμη. Απλά να σα υπενθυμίσω ότι στι Ιουλίου 9 Ιουλίου θα ε, ε, ψηφίσουμε. Είμαι σίγουρος ότι οι δύο εισηγητές θα συνεργαστούν με τους σκιώδους εισηγητές για να προγραμματίσουν, ε, για να προγραμματίσουν έναν κατάλογο ψηφοφορίας ε, πάρα πολύ δύσκολο, μοναδικά δύσκολο. Ελπίζω να τα καταφέρουμε. Ο κύριος Μάιρ θα είναι εδώ για να αποτελέσει μάρτυρα αυτού του φοβερού γεγονότος όταν γίνει και ελπίζω να έχουμε τη δυνατότητα να το, να το συζητήσουμε και στο πλαίσιο της ε, ψηφιακής αγοράς, ενιαίως ψηφιακής αγοράς ε, βλέπω ότι έχει μειωθεί το πεδίο ε, εφαρμογής ε, και αυτό έχει βέβαια σχέση με αυτό που ψηφίσαμε σήμερα το πρωί, μεγάλη σχέση μάλιστα. Υπάρχει μια πρόταση από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων ε, έδωσε μεγάλη σημασία σε αυτή τη γνωμοδότηση και μάλιστα εμείς την ψηφίσαμε εδώ με... και εγκρίθηκε με πολύ μικρή διαφορά. Ε, θα είναι λοιπόν πολύ ενδιαφέρουσα για τους ίδιους λόγους η ψηφοφορία στις 9 Ιουλίου γιατί άνθρωποι σε διαφορετικές πολιτικές ομάδες ε, έχουν διαφορετικές απόψεις. Ε, αυτό θα πει πολιτική. Ε, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ τους συνεισηγητές που συνεργαστήκατε τόσο πολύ παρά το γεγονός ότι διαφωνείτε μεταξύ σας. Άλλωστε αυτό θα πει πολιτική επαναλαμβάνω. Ελπίζω να απολαύσατε και όσοι μας παρακολουθείτε από το ίντερνετ αυτήν τη συζήτηση. Το απόγευμα έχουμε μία ακρόαση για την ασφάλεια του διαδικτύου, ε, για τη σχετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, έχουμε προσκεκλημένους ε, από τη Europol, από την Εστονία, διάφορους προσκεκλημένους. Σας καλούμε λοιπόν να παραστείτε στις 3 η ώρα μέχρι τις 5 για την ακρόασή μας και καλό βέβαια και το διαδικτυακό κοινό μας να μας παρακολουθήσει. Ευχαριστώ πολύ.